friends, please take your seats. Να καθίσετε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Θα ξεκινήσουμε με την ε, αποδοχή της ημερησίας διάταξης η οποία έχει ήδη διανεμηθεί. Έχουμε κάποια αιτήματα για τροποποιήσεις βέβαια. Ο εισηγητής της ερευνητικής αρμοδιότητας του Κοινοβουλίου, ο Ραμόν Χουαρέγγι, έχει ζητήσει το 6 για την άσκηση από πλευράς του Κοινοβουλίου του δικαιώματος του αυτού να συζητηθεί πριν από την ψηφοφορία έτσι ώστε να υπάρξει συζήτηση και να αποφασίσουν αν θέλουν τα μέλη να ψηφίσουν μια νέα εντολή για τις διαπραγματεύσεις. Στη τελευταία συνάντηση της ΑΦΚΟ η Επιτροπή δέχτηκε την πρόταση του εισηγητή να προετοιμάσει ένα έγγραφο εργασίες το οποίο θα κατατεθεί στη συνάντηση της 3ης Δεκεμβρίου μιας και το Συμβούλιο επιθυμεί να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις γύρω από το θέμα αυτό, η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου θα το συζητήσει το θέμα στη συνάντησή του την Παρασκευή 20 του μηνός. Δεύτερον, η κυρία Μπρέσο, η για την ετήσια έκθεση 14 για την προστασία των ε, ε, χρηματοπιστωτικών συμφερόντων της Ένωσης, ζήτησε το 7 να συζητηθεί επίσης πριν από την ψηφοφορία. Προτείνω λοιπόν το 6 και το 7 να τεθούν σε συζήτηση πριν από την ψηφοφορία και η ψηφοφορία να ακολουθήσει α, στις 10 η ώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ευχαριστώ κύριε Σόπφλιν. Όχι αντίρρηση. Θα ήθελα να καταγράψετε όμως μια κάποια δυσφορία από μέρους μου. Γιατί χθε το βράδυ άλλαξε η πρόταση για την ημερήσια διάταξη. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα σωστό. Τώρα που το εξηγήσατε έχει λογική αυτό το οποίο έγινε, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτή μια αλλαγή η οποία μπορεί να γίνεται την τελευταία στιγμή. Για το μέλλον λοιπόν παρακαλώ θα πρέπει να εμείνουμε στην εμερήσια διάταξη έτσι όπως έχει προαποφασιστεί μετά από διαπραγμάτευση. Και πριν ξεκινήσουμε ε, για την έκθεση Φουαρέγκουι, αλλά θα τα πω αυτά αργότερα. Θα επανέλθουμε λέει ο Πρόεδρος. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Κατανοώ πλήρως τη δυσκολία που δημιουργείται. Η αλλαγή έγινε Τη στιγμή που ενημερωθήκαμε για τα αιτήματα αυτά, αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα θα προσπαθήσουμε στο μέλλον να αποφεύγουμε τέτοιου είδους αλλαγές. Η κυρία Μπρέσο. Απλά να πω ότι εμείς το είχαμε ζητήσει εδώ και αρκετές ημέρες να γίνει η συζήτηση πριν. Ε, και γιατί χρειαζόμαστε περισσότερους παρόντες στην ψηφοφορία. Αυτό το αίτημα είχε σαν στόχο να οργανωθούμε με πιο σωστό τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ μπορώ να περιμένω, δεν έχω... Problem. Okay, well. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θα προσπαθήσουμε να αποφεύγουμε τέτοιες καταστάσεις στο μέλλον. Δεκτή λοιπόν η μερίσια διάταξη. Στις ανακοινώσεις του Προέδρου. Διακόπτει ο κύριος Σίλβα Περέιρα. Η κυρία Χούμπνερ θα κάνει τις ανακοινώσεις όταν έλθει αυτή. Οπότε δεν υπάρχουν ανακοινώσεις και περνάμε απευθείας στο σημείο 6. Πρόταση λοιπόν κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος έρευνας του Κοινοβουλίου. Θα δώσω το λόγο στον Ραμπόν Χουαρέγγι. έχει το λόγο. Oh, yes. Uh, ναι, συγγνώμη. Ο κύριος Σόφλιν ζήτησε το λόγο, παρακαλώ εσείς. Ευχαριστώ και πάλι, Πρόεδρε. Θα ήθελα να διαβιβάσω μια πληροφορία στον κύριο Χάουρεγγι. Εξ όσων γνωρίζω θα ζητήσετε την εντολή για να διαπραγματευτείτε με το Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ε, είναι σύμφωνο, αλλά ε, παρακαλούμε να συγκληθεί ε, συνεδρία των σχεδόν εισηγητών προηγουμένως, αν μπορείτε να το δεχτείτε. ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοδομητική παρέμβαση. Ο Ραμόν Χαουρίγκε. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Βιάζομαι να απαντήσω αμέσως στον κύριο Σόφσεν. Βεβαίως, αυτή την πρόθεση έχω. Φυσικά ως εισηγητής. Ανέκαθεν άλλωστε όταν είχαμε ε, διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα συγκαλούσαμε ε, συνεδρίαση των σχεδόν των μαζί μου πριν οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Επιτρέψτε μου λίγο να σας θυμίσω γιατί έχουμε ξανάρθει εδώ για αυτό το θέμα. Πάρα πολύ σύντομα, δεν θέλω να επεκταθώ για να σας εξηγήσω πώς έχει η κατάσταση. Θα θυμάστε ότι το Μάιο του 2012, στην προηγούμενη θητεία, το Κοινοβούλιο ενέκρινε για πρώτη φορά την έκθεση David Martin τότε. Ήταν το πρώτο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο για να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επί 1,5 χρόνο, από το 12 στο 14, οι διαπραγματεύσεις αυτές έγιναν με βάση τη συγκεκριμένη έκθεση. Μάρτιν, δεν υπήρξε τελική συμφωνία, κάποιες προσεγγίξεις σε ορισμένα επιμέρους θέματα, αλλά όχι οριστική συμφωνία. Η ΔΕ Επιτροπή μας συνταγματικών υποθέσεων αποφάσισε για να μην χαθεί η έκθεση ε, με το τέλος της θητείας αποφάσισε να την εγκρίνει ακριβώς μόνο για να μην ακυρωθεί. Και το 2014, τον Απρίλιο συγκεκριμένα, ενέκρινε το Κοινοβούλιο το κείμενο. Δυστυχώς αυτή η έγκριση έγινε παρά την επιστολή που είχαν απευθύνει στο Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου, Γενική Γραμματής ε, του Συμβουλίου και της Κομισιόν, όπου ε, ανέλυαν ε, όλες τους τις αντιρρήσεις τεκμηριωμένα, στοιχειοθετημένα, με νομικά επιχειρήματα που έλεγαν για ποιο λόγο ήταν απαράδεκτα κάποια ζητήματα και κάποιες ρυθμίσεις που παραβίαζαν τις συνθήκες ή την Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, αποφάσισε το Κοινοβούλιο να εκρίνει τον Απρίλιο του 2014 την έκθεση Μάρτιν, για να μην χαθεί. Τώρα, με την έναρξη της νέα θητείας, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ανέφερε σε μένα να ασχοληθώ με την υλοποίηση όλων αυτών. σα κατέθεσα το Γενάρη του 2015 ένα έγγραφο εργασία για να ξαναρχίσει διάλογο με τα θεσμικά όργανα. Από το κείμενο εκείνο του Ιανουαρίου, την κατάθεσή του και μετά δηλαδή, είχα διάφορες συζητήσεις με τη Λετωνική Προεδρία πρώτα, φυσικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια με τους διάφορους ε, σκιώδεις εισηγητές που από την αρχή συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια και μπήκαν στη διαπραγματευτική ομάδα. Πλην όμως δεν κατέστη δύνατο να επιτευχθεί εντολή στο Συμβούλιο για το διάλογο αυτό που στην αρχή ήταν διερευνητικός όσο και άτυπος. Εμείς δεν θέλαμε τίποτα άλλο, απλώ να βολιδοσκοπήσουμε ποιες ήταν οι δυσκολίες για να επαναλάβουμε τις επαφές και να δούμε τι δυνατότητες έχουμε να φέρουμε κοντά μας το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα διάλογο για να γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι τα προβλήματα και ποιες θα μπορούσαν ενδεχομένω να είναι και οι λύσει. Δυστυχώ, το Συμβούλιο ποτέ δεν έλαβε εντολή η πρώτερη έγκριση. Γιατί τώρα δεν ξέρω, είχε αναστέλουσες μειοψηφίες ή δεν υπήρχε επαρκή συνένεση. Πάντως, ε, όσες ε, συνεδριάσεις ε, έγιναν και συγκλήσεις, από όλες τις συνεδρίες που είχαν συγκληθεί, μία μόνο διεξήχθη τον Ιούνιο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απουσία του Συμβουλίου. το οποίο Συμβούλιο ευνηδιαστικά την παραμονή της συνεδρίασης και συγκεκριμένα η Λετωνική Προεδρία ακύρωσε την έλευσή του. Μέχρι το Σεπτέμβριο λοιπόν πρακτικά τράβηξαν έτσι τα πράγματα και εμφανίζεται η Προεδρία πλέον του Λουξεμβούργου. Θυμίζω ότι στην αρχή της θητείας τους εγώ ήμουν πάρα πολύ έντονος τη συνεδρίαση και έλεγα και ζητούσα να το λύσει αυτό το θέμα της έλλειψης επικοινωνίας η Λουξεμβουριανή Προεδρία. Στη συνέχεια το συζήτησα μαζί του και με το επιτελείο του. Υπήρχε μια έντονη ε, αλλαγή, ανταλλαγή επιστολών, αλληλογραφία για να δούμε πώς μπορεί να δοθεί εντολή διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο. Και έτσι έχουν σήμερα τα πράγματα. Οι δηλώσεις προθέσεων και η προθυμία του εισηγητού δεν είναι αρκετές για το Συμβούλιο, ούτε οι επιστολές της Προέδρου Χιούμπνερ. Το Συμβούλιο, για να το πω έτσι, ζητάει από την Επιτροπή μας ε, να δηλώσει ότι είναι πρόθυμοι να λυθούν οι νομικές δυσκολίες ε, που έλεγαν στην επιστολή τους το Απριλίου του 2014, πριν εγκρίνει η Ολομέλεια την έκθεση Μάρτιν. Επίσημα δηλαδή θέλει το Συμβούλιο να δηλώσει η Επιτροπή ΑΦΚΟ ότι προτίθεται να λύσει αυτά τα προβλήματα με νέες λύσεις. Διαφορετικές από ε, αυτές που είχαμε εγκρίνει στην έκθεση Μάρτιν. Κατά την άποψή μου είναι αναπόφευκτο κάτι τέτοιο. Γιατί δεν πρόκειται να έρθει ο λόγο κανονισμό αν δεν τα βρούμε με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίε και κύριοι. Ή θα συμφωνήσουμε με Συμβούλιο και Κομισιόν το νέο κείμενο το οποίο όμως θα είναι καινούριο σε κάποιους παραγράφους, όχι η έκθεση Μάρτιν, είτε θα καταρρεύσει. Διότι το άρθρο 226 της συνθήκης ορίζει ξεκάθαρα ότι η έγκριση του κανονισμού για το δικαίωμα στην έρευνα και στην εξέταση ζητεί, απαιτεί πρώτερη ε, συμφωνία του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η συμφωνία δεν υφίσταται. Τι να κάνουμε τώρα προβάλλουν νομικές αντιρρήσει και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά τη γνώμη μου ευσταθούν αυτά που λέγουν. Υπάρχει, γίνεται αυτή η νομική συζήτηση αλλά και πολιτική που είναι σημαντική για το θέμα αυτό. Διότι προφανώς το Κοινοβούλιο θέλει να εξασφαλίσει ότι οι εξεταστικέ επιτροπές θα έχουν σημαντικέ δυνατότητε για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά του. Σε κάθε κοινοβουλευτικό σύστημα εκφύσεως υπάρχουν τέτοιες επιτροπές, αλλά θα πρέπει να έχουν και τις δυνατότητες που χρειάζονται για να κάνουν τη δουλειά τους, την έρευνα και την εξέταση αυτή, που θα έχει αποφασίσει αρχικά το Κοινοβούλιο. Αλλά όπως σας είπα, αυτό που αποφασίσαμε προσκρούει σε διάφορα προβλήματα, εμπόδια. Ας πούμε, όταν κάτι εκκρεμεί στη δικαιοσύνη ενός κράτους μέλους, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει έρευνες στα έγγραφα, είναι πιστευτικά διαβαθμισμένα ή κατά πόσο μπορεί το Κοινοβούλιο να αναγκάζει μάρτυρες να έρθουν να καταθέσουν, να επιβάλλει κυρώσεις σε περίπτωση που αυτοί αρνούνται. Είναι 5-6 τα προβλήματα σε ένα σύντομο κατά τα άλλα κείμενο. Δεν είναι πάνω από 20 άρθρα, παρόλα αυτά υπάρχουν προβλήματα. Και ζητούν μια νέα συνένεση. Όχι ακριβώς νέα, δεν υπήρχε παλιά ποτέ συνένεση. Μια συνένεση τελεία. Σκέτη. Πιστέψτε με κυρίε και κύριοι, το έγγραφο που καταθέτω αυτή τη στιγμή είναι τελευταία ευκαιρία που έχουμε έτσι ώστε το Συμβούλιο να αναθεωρήσει τη θέση του και να δεχτεί την έναρξη επισήμων τυπικών διαπραγματεύσεων. Αν μου επιτρέπετε και ένα σχόλιο. Αυτό είναι το κλειδί που ανοίγει την πόρτα του κάστρου, αν θέλουμε έτσι να το χαρακτηρίσουμε και το χρειαζόμαστε αυτό το κείμενο. Σας ζητώ την εμπιστοσύνη σας. Το κείμενο αυτό μπορεί να το δεχτεί το Συμβούλιο ως βάση πολιτικής βούλησης και έκφρασης προθυμίας της Επιτροπής μας για να επιτευχθεί αυτή η απαραίτητη συνένεση. Σε περίπτωση λοιπόν που δοθεί εντολή στο Συμβούλιο για διαπραγμάτευση με το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έτσι κι αλλιώς αυτοί θέλουν να διαπραγματευτούν, θα ε, είναι το κλειδί για να αρχίσουν οι επίσημε διαπραγματεύσει. Απαντώ και πάλι στον κύριο Σόφλιν και στον κύριο Βίλαντ που εχθέ το βράδυ, ο σκιώδη ηγητή του ΕΛΚ, που είπε ότι θέλει να έχουμε συνεννόηση μεταξύ μα προηγούμενη βεβαίω, αλίμονο. σας λέω να συμφωνήσουμε για αυτό το κείμενο και μόλις μας δηλώσει το Συμβούλιο ότι επιτέλους έχει εντολή, διαπραγματεύσεις θα κάνει μια ομάδα δική μας που θα είναι όλων των συντονιστών και όλων των ομάδων, των, συγγνώμη, των σκιωδών εισαγητών Θα συνεννοηθούμε βεβαίως και με την πρόεδρο Χιούμπνερ και με την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Και βάσει του άρθρου 73 του κανονισμού η πρόεδρός μας θα ορίσει τη διαπραγματευτική εντολή επίσημα. Εξ ονόμα της Επιτροπής. Είναι απαραίτητο αυτό το βήμα, συνάδελφοι, και τελειώνω λέγοντας το εξής. Σε περίπτωση που δεν λυθεί έτσι το πρόβλημα θα πρέπει να επανέλθουμε εδώ να το συζητήσουμε με όλους τους συντονιστές και την πρόεδρο Χιούμπνε για να ανεβάσουμε αυτό το θέμα, αυτή τη σύγκρουση σε επίσημο, ανώτερο επίπεδο και να υπάρχει επίσημη διοργανική ε, σύγκρουση. Εμείς έχουμε εντολή ε, από τις συνθήκες για να νομοθετούμε και θα πρέπει να την ασκήσουμε. Αν δεν υπάρχει βούληση από την άλλη πλευρά, η δική μας Επιτροπή εδώ, ΑΦΚΟ και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να το φέρουν σε ανώτατο επίπεδο αυτό το θέμα, αυτή την κόντρα. Αυτό είναι κάτι την περίπτωση. Ούτε το προβλέπω, ούτε το επιθυμώ. Αλλά αυτό που σας προτείνουμε είναι το απαραίτητο εκείνο βήμα για να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Και το Γενάρη να έχουμε, ελπίζω, επίσημη διαπραγμάτευση. Η δική μας ομάδα να είναι όλοι οι σκιώδεις όλων των ομάδων και από την άλλη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβούλιο. Και φυσικά πάντα και με την Πρόεδρο Χιούμπνερ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι σαφής η πρόταση. Κύριε Σόπφλη, να είστε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, σύντομος θα είμαι. Πιστεύω πως έγινε εξαιρετική δουλειά, διότι υπάρχει το θεματολόγιο, υπάρχει το τι πρέπει να κάνουμε και είναι σαφές αυτό. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός φάκελος και ένας πάρα πολύ δύσκολος επίσης. Και μου φαίνεται ότι αυτή η πολυπλοκότητα απορρέει από το ότι αυτό είναι το σημείο στο οποίο συναντάται ο νόμος με την πολιτική. Και εγώ θα έλεγα ότι το κοινοβούλιο το αφορά αυτό το θέμα. Έχει να κάνει με τη ε, δύναμη εκπροσώπησης των πολιτών του και το δικαίωμα έρευνας λοιπόν. Επίσης θα ήθελα να πω ότι και για τα άλλα θεσμικά όργανα υπάρχουν κάποιες ευαισθησίες, κρατικές ευαισθησίες. Και είναι ένα θέμα το οποίο ίσως θα έπρεπε να εξετάσουμε μέσω μιας εξεταστικής επιτροπής κάποιου, κάποιου κράτους μέλους. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν υπόψη όλες αυτές οι ιδιαιτερότητες που κάνουν το ζήτημα αρκετά περίπλοκο. Και πιστεύω πως επίσης είναι καιρός να προχωρήσουμε με αυτό το θέμα. Το θυμάμαι και από προηγούμενες κοινοβουλευτικές θητείες. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πόσο ε, καιρό ασχολούμαστε με αυτό. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι πάντως με την δουλειά που έχετε κάνει και θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή τύχη στις διαπραγματεύσεις σας με τα άλλα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπρέσο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και από τη δική μας πλευρά θα συμφωνήσουμε με τη διαδικασία την οποία προτείνει ο συνάδελφος Χαουρέγγι. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να δώσουμε μια σωστή εντολή στον διαπραγματευτή και να ενημερώνει ε, πλήρως όλες τις πολιτικές ομάδες μέσω των συντονιστών ή μέσω των σκιωδών όπως αυτό το προτιμά και μετά ελπίζω να πετύχουμε, εν πάση περιπτώσει, ένα αποτέλεσμα ικανοποιητικό. Δεν υπάρχει νομίζω άλλη λύση από το να αποδεχθούμε την διαπραγμάτευση. Εμείς συνεχίζουμε να έχουμε την εντολή και έχει σημασία να καθορίσουμε ένα ακείμενο συμφωνημένο Μπορεί να αφήσουμε λίγα φτερά στο πορεία, αλλά παρόλα αυτά θα καταλήξουμε σε μια κάποια λύση. Εγώ έχω πλήρη εμπιστοσύνη στις διαπραγματευτικές δυνότητες του Ραμών και να προχωρήσουμε. Το θέμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ή θα συμφωνήσουμε και εμείς λοιπόν με τις προτάσεις ε, του Χάουρεγγι και του ευχόμεθα καλή τύχη έτσι ώστε να πετύχουμε τους στόχους τους οποίους όλοι έχουμε. Γνωρίζω τον κύριο Χάριγκ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι νομίζω ικανός να εργαστεί σε ένα τόσο δύσκολο περιβάλλον. Θα υπάρξουν πάρα πολλές δυσκολίες, υπάρχουν όμως και θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, στα οποία εμένουμε εμείς στο Κοινοβούλιο και ελπίζω ότι θα το πετύχουμε. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλο το λόγο, οπότε θα επανέλθουμε την ώρα της ψηφορίας στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ραμόν, α. Τίποτα, μόνο να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη και ελπίζω να μην τους απογοητεύσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παίρναμε τώρα στο σημείο 7 της ημερησίας διάταξης με τη έκθεση για το 2014 για την καταπολέμηση της απάτης και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαρισέντες Μπρέσο για να μας παρουσιάσει τη θέση της σχετικά με τις τροπολογίες που έλαβε. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα κάνω μια πλήρη παρουσίαση του εγγράφου, διότι ήδη το παρουσίασα στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ε, για εμένα ως εισηγήτρια κάποια θέματα είναι ιδιαίτερη σημασία και θα σας τα αναφέρω αμέσως. Καταρχάς, ε, η, ε, ξεκάθαρη, ένας διαχωρισμός ανάμεσα στην απάτη και στο σφάλμα, η βελτίωση της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο οριζόντιος ε, χαρακτήρας των ε, πολιτικών. Σύμφωνα με το άρθρο 325 της Συνθήκης. Υπάρχουν 28 τροπολογίες, μπορώ να δεχτώ τις 18 από αυτές και θα προτείνω δύο συμβαστικές τροπολογίες που θα συμπεριλαμβάνουν 6-7 περίπου από τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν. Θα ήθελα να τονίσω ότι κατέβαλα ιδιαίτερε προσπάθειες για ε, τις ε, τροπολογίες σε αρκετά θέματα. Καταρχάς ε, για την περισσότερη διαφάνεια στην διαδικασία, τον, την διαφάνεια του, των ευρωπαϊκών κονδυλίων που χρησιμοποιούνται και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο για και την σύσταση μίας υπηρεσίας κατά της απάτης έπειτα για την ε, διαφάνεια των ε, δημοσιοσυμβάσεων, για το άρθρο 14 για παράδειγμα σχετικά με αυτό, η τροπολογία 12 είναι η σχετική, έπειτα για την επιτάχυνση της διαδικασίας ε, υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που είναι ένα πολύ περίπλοκο θέμα και βλήθηκαν πολλές τροπολογίες γι' αυτό. Έχω προτείνει λοιπόν εδώ μια συμβαστική τροπολογία η οποία θα συμπεριλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερες ε, τροπολογίες. Και τέλος η δημοσίευση της αξιολόγησης των συμφωνιών με τις εταιρείες ε, καπνού. Δεν βλέπω τώρα κάποιους άλλους ε, προβληματικούς τομείς στην ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σόπφλιν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την κυρία Μπρέσο για την δουλειά που έκανε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Υπάρχουν σίγουρα δυσκολίες, όμως βλέπω ότι τις έχετε αντιμετωπίσει και τις έχετε επιλύσει ικανοποιητικά. Πιστεύω πως η πρότασή σας ε, είναι κέρια σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πιστεύω πως ε, όντως δημιουργείται θέμα εθνικών αρμοδιοτήτων και θα τοποθετηθούμε από αυτού. Σχετικά με την ανεξαρτησία και την διαφάνεια, ε, να πω ότι συμφωνώ μαζί σας, είναι όντως ζωτική σημασία το θέμα αυτό και πρέπει να εργαστούμε εντατικότατα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για όλη τη δουλειά που κάνατε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντουράν, έχετε το λόγο. Σύντομα πρόεδρε. Ήδη αναφερθήκαμε σε αυτό την τελευταία φορά. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μπρέσο. Έχουν υπάρξει βήματα ικανοποιητικά και οι παρατηρήσεις τις οποίες έκανα στην τελευταία συνάντηση βλέπω ότι επέτρεψαν να γίνουν κάποια βήματα προς την κατεύθυνση των θέσεών μας. Δεν είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την Επιτροπή Εποπτείας της ΣΟΛΑΦ. Καταλαβαίνω ότι είναι περίπλοκο το θέμα, ιδιαίτερα στο δημοσιονομικό κομμάτι. Δεν μπορώ να επιμείνω πλέον, αλλά νιώθω μια κάποια δυστημία. Για τα υπόλοιπα τώρα, τίθεται και το θέμα του δίκτυ διαφθοράς ο δείκτης διαφοράς ε, είναι σαν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δίνει δείκτες ε, για το ποσοστό απορρόφησης των οδηγιών στις διάφορες χώρες. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε να κάνει κάτι τέτοιο η Επιτροπή για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της διαφθοράς και να μπορέσει να δώσει κάποιες ε, προτάσεις για την αντιμετώπιση τους. Ίσως είναι κάτι που θα πρέπει να ψάξουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ την Μεσεντές για την προσπάθειά της. Και εμείς συμφωνούμε και συγχαίρουμε την κυρία Μπρέσο. Είναι επεξεργασμένες οι θέσεις της και μπορούμε να τη στηρίξουμε είναι βασικό το θέμα και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα και για τη δική μου χώρα και τον λαό μου. Τελικά σχόλια από τη Μεσέντες. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους πήραν το λόγο μέχρι τώρα. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για τα θέματα που βρίσκονται σε κρεμότητα. Να πω στον συνάδελφο Ντουράν ότι εγώ είμαι επιφυλακτική σε σχέση με τους λεγόμενους σύνθετους δείκτες. Ένας δείκτης διαφθοράς σε διάφορες χώρες που να αποτελείται από πολλά συστατικά διαφορετικά μεταξύ τους είναι δύσκολο να οδηγηθούμε σε μια σωστή ε, θα έλεγα στάθμιση. Ξέρετε οι δείκτες ας πούμε για τις δραστηριότητες των βουλευτών. Ε, ξέρετε ότι μας εκπλήσουν αυτό γιατί κάποιοι που κάνουν λίγα πράγματα φαίνεται σαν να έχουν κάνει πολλά. Είμαι λοιπόν επιφυλακτικός σε σχέση με τέτοιου είδους δείκτες που μπορεί να οδηγεί σε αποτελέσματα όχι ιδιαίτερα χρήσιμα, σε αποτελέσματα που κινδυνεύουν να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα παρά λύσεις. Πάντως θα το σκεφτούμε το θέμα και εγώ και οι συνάδελφοι μήπως βρούμε μία λύση διαφορετική έτσι ώστε να το μελετήσουμε εκ νέου γιατί πριν προτείνουμε έναν τέτοιο δίκτυ νομίζω ότι θα είχαμε και εμείς ε, το συμφέρον, κάθε συμφέρον ε, να είμαστε επιφυλακτικοί. Είναι δύσκολο ε, να ανακατεύει κανείς εντελώς ετερόκλητα πράγματα και να θέλει να βγάλει συμπεράσματα από αυτό. Τα μήλα και τα αχλάδια λένε στα γαλλικά, αλλά υπάρχουν και χειρότερα μεταξύ τους εντελώς ασύμβετα και ε, α, πράγματα τα οποία δεν συγκρίνονται. Ξέρω ότι κάποιοι δείκτες και στον κοινωνικό τομέα δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Δεν είμαι λοιπόν ε, καταρχήν κατά, αλλά έχω αμφιβολίες για τη χρησιμότητα. Θα συζητήσω το θέμα με τον κύριο Ντυρό ο οποίος έχει προτείνει τη συγκεκριμένη τροπολογία. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε λοιπόν και το θέμα αυτό. Θα δώσω τώρα το λόγο στην πρόεδρό μας, η οποία μόλις αφήσει και μπορεί να κάνει τις ανακοινώσεις. I'm sorry, we just Είχα μια συνάντηση με το Κορεπέρ για τον εκλογικό νόμο. Να σας ενημερώσω λοιπόν για τις αποφάσεις των συντονιστών την 29η Δεκάτου σχετικά με τους διορισμούς. Οι συντονιστές αποφάσισαν να διορίσουν τον κύριο Ατόντο σαν εισηγητή για την έκθεση πρωτοβουλίας για την ηλεκτρονική δημοκρατία. Τον κύριο Ντιό από τους Πρασίνους είναι εισηγητής για τη γνωμοδότηση της ΑΦΚΟ στην έκθεση της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου για την Απαλλαγή 2014 Γενικός Προϋπολογισμός με Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του προϋπολογισμού στο 14. Το ΕΛΚ παίρνει και θα μας πει ποιος είναι ο εισηγητής για τη γνωμοδότηση της ΑΦΚΟ, για την έκθεση της ΛΥΜΠΕ, για την έκθεση επίσης του 2014 για την εφαρμογή της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Σχετικά τώρα με την έκθεση, την οποία ζητήσαμε να αναλάβουμε στην Επιτροπή των Προέδρων εδώ και αρκετό καιρό, και υπήρξε πρόταση για αλλαγή τίτλου. Σχετικά με την έκθεση αυτή, οι συντονιστές είπαν ότι θα πρέπει να διατηρηθεί ο παρόν τίτλος και ζήτησαν από την Πρόεδρο να υποβάλει την έκθεση προς έγκριση στην διάσκεψη των Προέδρων. Ε, και η ΕΚΟΝ επίσης θα είναι συνδεδεμένη επιτροπή σχετικά με το υπόλογο το δημοκρατικό και την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Πήραμε επίσης επιστολές από τον πρόεδρο Αλάλα Μασούρ της Επιτροπής Τάξα για τη μη συνεργάσιμη στάση ορισμένων πολυεθνικών επιχειρήσεων στα πλαίσια των εργασιών της Επιτροπής του για τα λεγόμενα tax rulings. Και αποφασίσαμε στη συνάντηση των συντονιστών ότι οι επιστολές αυτές περιλαμβάνουν κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί στα πλαίσια ε, των πιθανών αλλαγών των κανόνων των διαδικαστικών λειτουργίας των ειδικών επιτροπών. Οι συντονιστές είπαν επίσης ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και στα πλαίσια της εκθέσεως Giggold για τη διαφάνεια ε, των ευρωπαϊκών οργάνων. Είπαμε ότι θα πρέπει να ενημερώσουμε και το Φερχόστατ για το θέμα, έτσι ώστε να δει αν είναι δυνατόν τέτοιου είδους θέματα να αντιμετωπιστούν και στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων της νέας διοργανικής συμφωνίας για καλύτερη νομοθετική δραστηριότητα. Σχετικά τώρα με τις προτάσεις ε, ψηφισμάτων, οι συστάσεις των συντονιστών είναι οι εξής. Για το πρώτο που αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο και το δημοψήφισμα για την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρούμε ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια μιας έκθεσης κανονικής της ΑΦΚΟ. Η συγητής μας είναι ο κύριος Φερχόφστας πιθανές εξελίξεις για την παρούσα θεσμική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, για τις δαπάνες για πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπαμε ότι δεν θα υπάρξει από πλευρά μας μια αυτόνομη πρόταση, αλλά η πρόταση αυτή θα αποσταλεί στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών για πιθανή εξέταση από πλευράς της στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Τώρα, για τις διακρίσεις εις βάρος των μη εγγεγραμμένων μελών. Αυτό θα απασχολήσει την ομάδα εργασίας για τον κανονισμό και το ψήφισμα τώρα για τη μεγαλύτερη διαφάνεια στα ευρωπαϊκά όργανα δεν θα υπάρξει συνέχεια από πλευρά μας και πήραμε την απόφαση έτσι και αλλιώς το θέμα αυτό να συμπεριληφθεί πάλι στην έκθεση Giggold. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχουν αγκυρίσεις σε σχέση με τις συστάσεις αυτές των συντονιστών, θεωρώ ότι γίνονται δεκτές από την Επιτροπή μας. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σχετικά με την προγραμματισμένη επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Κοινοτήτων, εμείς προβλέπουμε να οργανώσουμε την επίσκεψη αυτή ε, στις 27-28 Ιανουαρίου του 2016 και θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως για τις τελικές ρυθμίσεις. Τώρα θα πρέπει να περιμένουμε να φτάσουμε στην ώρα της ψηφοφορίας στις 10. Λοιπόν, για 5-6 λεπτά διακόπτουμε. Dear colleagues, I would like to start Αγαπητοί συνάδελφοι, ας αρχίσουμε την ψηφοφορία. Έχουμε τρία θέματα για την διαδικασία της ψηφοφορίας. Το πρώτο έχει να κάνει με την ψηφοφορία, με αυτό που συζητήσαμε νωρίτερα, ε, την εξεφύρα Ραμόν Χαουρέγγι και να σας πω πως η ψηφοφορία για τον πολιτικό προσανατολισμό του εγγράφου εργασίας, στο οποίο επιβεβαιώνεται από την Επιτροπή μας η πρόθεση ε, να ασχοληθούμε με τις ε, ανησυχίες που ανέφερε το Συμβούλιο και με την ε, εντολή που θα δώσουμε στον εισηγητή για να συνεχίσει τις επαφές με το Συμβούλιο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, σε αυτό το στάδιο, αλλά και στην Επιτροπή για να συνεχίσει τι ενέργειε για την έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων. Και επίσης να σας ενημερώσω ξανά ότι οι επίσημε διαπραγματεύσεις θα γίνουν μετά από την ε, σύσταση της επίσημης διαπραγματευτικής ομάδας. Μόλις δηλαδή έχουμε την επιβεβαίωση από το Συμβούλιο, θα αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω εάν εγκρίνεται την πρόταση αυτή. Είστε σκορπισμένοι, δεν είναι κανείς στη μέση. Ποιος είναι υπέρ λοιπόν αυτής της πρότασης να στηρίξουμε τον Ραμόν Χαουρέγγι. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Κανένας. Ραμόν λοιπόν, πήρες ό,τι μας ζήτησες. Περνάμε τώρα στο δεύτερο σημείο της ε, μερίσας διάταξης για την ψηφοφορία, μια γνωμοδότηση του Παύλου Ραντζέλ για τον ρόλο των θεσμικών οργάνων. Okay. Can we... Can we start... Στο πλαίσιο των διεθνών, των και χρηματικών πιστοτικών, ρυθμιστικών οργάνων και φορέων. Ποιος είναι... Συμβαστική Α, ποιο είναι υπέρ. Ποιο είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά ηλεκτρονικός έλεγχος. Νομίζω πως ε, αλλά θα το κοιτάξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς. πέρα Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. δεν είμαι σίγουρη, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για το πρώτο μέρος. Πέρας ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε επίσης ηλεκτρονικά το δεύτερο μέρος της τροπολογίας. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Σ. Υπέρ. Με συγχωρείτε, λέει πρόεδρος. Είναι ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα της συμβιβαστικής Σ. είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται.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 Αποχές απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 25. Πέρας ψηφοφορίας. Τι έγινε. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίθηκε, αλλά ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ε, με 9 ψήφους υπέρ εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 8 ψήφους υπέρ 7 κατά. 28. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Ι e. υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται με νέα ψήφους υπέρ 7 κατά. 42 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 44 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος γιατί είναι 44 για το πρώτο τμήμα. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Καταπίπτει το δεύτερο τμήμα. Και περνάμε στην 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 47. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 47. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 49. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 50. Υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 50. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 9 ψήφι υπέρ, 9 κατά. Απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 13 ψήφους υπέρ, 3 κατά, 2 αποχές. Συγχαρητήρια Πάουλο. Τώρα θα ήθελα να σας πληροφορήσω πως ε, είχαμε την ψηφοφορία και την, τον κατεξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής όσον αφορά το περιεχόμενο και τη λειτουργία του Μητρώου για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα. Υπήρχε μια προθεσμή για τη διατύπωση ενστάσεων η πρόταση ενσύσταση για πρώιμη μη διατύπωση ενστάσεων από τους βουλευτές. Σύμφωνα με τον κανόνα 105, η προθεσμία έληξε στις 29 Οκτωβρίου, δεν υπήρξαν ενστάσεις, δεν υπήρχε κάποιο αίτημα παράτασης. Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή Αύκο Αύκο δεν θα υποβάλει πρόταση ψηφίσματος για το θέμα αυτό. Όμως Επαναλαμβάνω ότι οι πολιτικές ομάδες θα έχουν την ε, δυνατότητα να παρουσιάσουν την ε, ένστασή τους στην Ολομέλεια. Γι' αυτό λοιπόν τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες και πρέπει δυστυχώς να κάνουμε και ένα άλλο διάλειμμα διότι τελειώσαμε γρήγορα τις ψηφοφορίες. Θα αρχίσει λοιπόν η συνεδρίαση με τα Εθνικά Κοινοβούλια στις 10.30 Γι' αυτό λοιπόν διακόπτουμε την συνεδρίαση μέχρι τις 10.30. <laughs> Εσύ,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

Πάλι, dear Αγαπητοί συνάδελφοι, θα σας παρακαλούσα Normally people who... να καθίσετε. Τώρα συνήθω αυτοί που έχουν ιδιωτικές συνομιλίες δεν φορούν ακουστικά και δεν μας ακούνε. Οπότε πώς να τους κάνουμε να καθίσουμε. Σας ε, καλωσορίζω θερμότατα. Χαίρομαι πάρα πολύ διότι ξεκινάει εδώ μια νέα ε, παράδοση στην Επιτροπή μας μου είπαν ότι στο παρελθόν δεν υπήρχε τέτοια παράδοση συναντήσεων με εθνικά κοινοβούλια. Ε, είμαστε πολύ υπερήφανοι που καταφέραμε να συνενέσετε και να δεχτείτε την πρόσκλησή μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ έως ήρθατε από τα Εθνικά Κοινοβούλια, 13 τον αριθμό νομίζω είναι παρόντα, Εθνικά Κοινοβούλια. Θέλω να καλωσορίσω τον Μάρκ Άντζελ που είναι ε, της ε, Προεδρίας, εδώ εκπροσωπεί την Προεδρία, αλλά στο ε, Κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου προεδρεύει στην Επιτροπή Εξωτερικών Άμυνας, ε, Συνεργασίας Μετανάστευσης και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στη Βουλή των ε, αντιπροσώπων και θέλω να καλωσορίσω και τον Υπουργό Νικολά Σμιτ ε, που είναι Υπουργός Προεδρεύων. Έχετε αρχίσει να καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά τελειώνει η σκληρή δουλειά της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας, αλλά μια που είστε παρόν θα εκμεταλλευτούμε την Προεδρία μέχρι τελικής ε, πτώσεως. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Θέλουμε να καλωσορίσουμε και τον πρώτο Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξέφρασε την επιθυμία του να έρθει, αλλά δυστυχώ χτες το βράδυ τον κάλεσαν εκτάκτος στην Άγκυρα για μια συνεδρίαση τον κύριο Τίμερμανς. Όπως γνωρίζετε είναι πολύ κρίσιμη η περίοδος αυτή. Ε, γίνονται διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και τουρκικής κυβέρνησης και ε, αναγκάστηκε να μεταβεί στην Άγκυρα, αλλά έχουμε τον κύριο Πασκάλ Ντίνη, Διευθυντή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που εκπροσωπεί τον πρώτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Τίμερμαν. Δεν θέλω να καλωσορίσω άλλους, γιατί πάντα κάποιον θα ξεχάσω. Σας καλωσορίζω όλους λοιπόν συλλογικά και θα ήθελα να αναφέρω τους Τούρκους και Νορβηγούς συναδέλφους που έχουμε ενώπιόν μας από τα αντίστοιχα κοινοβούλια και με μεγάλη χαρά ε, σας καλωσορίζω εδώ. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι λάβαμε από τον Λόρδο Μπόσουελ, ε, τον πρόεδρο της ε, Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στη Βουλή των Λόρδων, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε λάβει μια επιστολή όπου εκφράζει την ανησυχία του ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που έχουμε ε, στην πρώτη ενότητα λέγει θα πρέπει να συζητήσουμε και το θέμα του διακυβολιστικού ελέγχου των ευρωπαϊκών οργανισμών. Ε, με χαρά λοιπόν θα ακούσουμε ό,τι έχετε να πείτε, αν θέλετε να επεκταθούμε και πέραν των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και να μιλήσουμε και για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς ε, ε, agencies, βεβαίω εφόσον υπάρχει τέτοια ανάγκη. Λάβαμε επίσης και μια άλλη πρόταση του Λόρδου Τιμ Πόσουελ που έχει κυκλοφορήσει, έχει δανειμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες. από την τριμερή συνεδρίαση των μελών της Βουλής, των Λόρδων της Βουλής των Κοινοτήτων και ε, των ε, ε, Βρετανών Ευρωβουλευτών. Στις 5 Νοεμβρίου συνεδρίασαν και έχουν κάνει ένα έγγραφο που ήθελα να μοιραστούμε και εμείς μαζί τους. Γιατί συνεδριάζουμε σήμερα, θα το γνωρίζετε φαντάζομαι όλοι σας, διότι ζούμε πολύ δύσκολους καιρούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ως βουλευτές εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κοιτάμε και το μέλλον. Έχουμε μικρές μάχες καθημερινές ή μεγάλες, πολύ σημαντικές, αλλά θα πρέπει να κοιτάμε και ένα ορίζοντα για το θεσμικό μας πλαίσιο και σε ποιο βαθμό μπορούμε να ανταποκρινόμαστε σε όλες αυτές τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Θα ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε μαζί την έκθεση της κυρίας Μερσέντες Μπρέσο και του κυρίου Μπροκ για τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας πλήρως το δυναμικό της συνθήκης της Λισαβόνας. Επίσης την έκθεση Γκί Φερχόφστατ που ε, προετοιμάζει ε, στην Επιτροπή μας για την ε, μελλοντική εξέλιξη. Όλα αυτά συνδέονται με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολλές και μεταξύ άλλων υπάρχει και ανάγκη να δούμε ποια είναι τα θεσμικά εργαλεία που έχουμε, η αρχιτεκτονική και η δυνατότητα διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όχι μόνο την αποτελεσματικότητα αλλά και τη δημοκρατική νομιμότητα και τη λογοδοσία των ευρωπαϊκών οργάνων λήψης αποφάσεων. Λοιπόν, δύο ενότητες έχουμε. Το πρωί θα συζητήσουμε τη μετεξέλιξη της θεσμική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το δεύτερο είναι το απόγευμα, η δεύτερη ενότητα, ε, μια ακρόαση ε, για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί της εκτελεστικής εξουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας αρχίσουμε λοιπόν, θέλω να δώσω μέσα στο λόγο σε τρεις εκπροσώπους. Τώρα την χάνει να είναι τρεις άνδρες. Στο κοινοβούλιο μας ε, αυτό μας λυπεί. Ε, να έχουμε μόνο άνδρες δηλαδή εδώ στο πάνελ, τι να κάνουμε, εκπροσωπούν τα θεσμικά του όργανα. Ο Μάρκ Άντζελ, εξ ονόματο λοιπόν τη Προεδρία του Λουξεμβούργου και ε, των Κοινοβουλίων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει το λόγο, Μάρκ. Ελπίζουμε οι βασικοί ομιλητέ να περιοριστούν σε ένα δεκάλεπτο και μόλις λήξει θα σας το επισημάνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Ντανούτα, αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Όπως ανέφερε και η Πρόεδρος, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα σημείο καμπής, διότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι μεγάλες. Ο διακοινοβουλευτικός διάλογος είναι αναγκαίος έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικότητα αυτές τις προκλήσεις. Γι' αυτό λοιπόν Χαίρομαι πολύ που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να συμπεριλάβει τα εθνικά κοινοβούλια σε αυτόν τον πολιτικό διάλογο. Υπάρχει και το έγγραφο εργασία τη ε, κυρία Εμπρέσου και του κυρίου Μπρόκ σχετικά με αυτό υπάρχει και μια νέα ε, διοργανική συμφωνία για καλύτερη νομοθεσία που αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση. Είναι αναγκαίος αυτός ο πολιτικός διάλογος για δύο λόγους. Καταρχάς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια αντιμετωπίζουν το γεγονός ότι οι αλλαγές στι συνθήκε δεν φαίνεται να είναι δυνατόν να γίνει στο άμεσο μέλλον. Κατα... Ε, έπειτα, Χρειάζεται βελτίωση της λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών και της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Έπειτα, πιστεύω πως μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι ο ρόλος ε, και η συμμετοχή των εθνικών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να ενισχυθεί. Πρέπει να ενισχυθεί σύντομα, το συντομότερο δυνατόν. Γι' αυτό λοιπόν ο πολιτικός ε, διάλογος ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι πιο σημαντικός από ποτέ. Πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας για τον καλύτερο έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας και σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Συμβουλίου. Ε, φυσικά δεν πρέπει να γίνει ε, σύγχυση και επικάλυψη αρμοδιοτήτων. Αυτές είναι προκλήσεις που έχουμε, αλλά ταυτόχρονα και ευκαιρίες συνεργασίας ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και θα ήθελα να σταθώ σε αυτό συγκεκριμένα σήμερα, διότι είμαι πεπισμένο ότι η συνεργασία ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με περισσότερη νομιμότητα. Δεν ήμουν ποτέ πιο σίγουρος ε, για το ότι υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται να έρθουμε πιο κοντά στους πολίτες και γι' αυτό χρειαζόμαστε τα Εθνικά Κοινοβούλια. Γι' αυτόν τον λόγο επίσης χρειάζεται καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ε, η κοινοβουλευτική διάσταση της Προεδρίας του Λουξεμβούργου προσπαθεί να ε, ασχοληθεί με την ενεργό συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων στα ευρωπαϊκά ζητήματα και είχαμε καλά αποτελέσματα. Ε, τα Εθνικά Κοινοβούλια, επίσης, μην ξεχνάτε, πως παίρνουν πολύ σοβαρά τον θεσμικό του ρόλο στα ευρωπαϊκά ζητήματα και η Προεδρία του Λουξεμβούργου προσπαθεί να εμβαθύνει το πολιτικό διάλογο και να ενισχύσει το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων σχετικά με την επικουρικότητα. Υπό την Προεδρία μου είχαμε δύο συνεδριάσεις της ΕΚΟΣΑΚ τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο όπου ασχοληθήκαμε με συνταγματικά ζητήματα. Είχαμε την ομάδα για τις κίτρινες και τις πράσινες κάρτες. Η τρίτη συνεδρίαση της ΚΟΣΑΚ σε λιγότερο από μία εβδομάδα θα ασχοληθεί επίσης με αυτά τα συνταγματικά ζητήματα και χαίρομαι πάρα πολύ ότι ο εσωτερικός κανονισμός ε, για το άρθρο 13 για την χρηστή ε, ε, διακυβέρνηση εγκρίθηκε υπό την Προεδρία μας. Τώρα, η διαδικασία της κίτρινης κάρτας στις δύο συνεδριάσεις ΚΟΣΑΚΑ έδειξε ότι χρειάζεται βελτίωση χωρίς αλλαγή συνθήκης. Επιπλέον, είμαι πεπισμένο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει τι προσπάθειέ τη για να διασφαλίσει την καλύτερη ποιότητα και την ε, ταχύτερη ε, απάντηση στις, ε, στα σχόλια και στι ερωτήσει των Εθνικών Κοινοβουλίων. Τώρα, όσον αφορά τον ενισχυμένο πολιτικό διάλογο, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε με ευελιξία σε σχέση με τα διαδικαστικά ζητήματα. Και αναφέρομαι στην πρόταση για νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία να σας αναφέρω κάποια σημεία τα οποία αφορούν την πράσινη κάρτα και έχουμε ήδη θέσει σε ισχύ. Πρώτη πρόταση, Τίμωθη Μπόσουελ από τη Βουλή των Λόρδων, ο οποίος ε, ασχολείται με τα ε, απόβλητα των τροφίμων, με την εσπατάλη των ε, τροφίμων και η απάντηση τη Επιτροπής έφτασε μόλις πριν από δύο μέρες. Η δεύτερη πρόταση από τους Λετωνού συναδέλφους αφορά την πράσινη κάρτα και την οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα. Και η τρίτη ε, πρόταση για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων παρουσιάστηκε πριν από μερικέ εβδομάδες στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση και τώρα θα ε, τεθεί πονάλης από τα εθνικά κοινοβούλια. Χρειάζεται λοιπόν ένα ελάχιστο όριο και μία ε, προθεσμία για την πράσινη κάρτα. Αυτά θα τα συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα στη συνεδρίαση της ΚΟΣΑΚ στο Λουξεμβούργο. Να σας υπενθυμίσω ότι ε, στα πλαίσια της διαδικασία της πράσινης κάρτας θα ήταν ευκταία η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσο το δυνατόν περισσότερο. Και σύμφωνα με το άρθρο 225 της συνθήκης, το δικαίωμα ε, να ζητηθεί από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση υπάρχει. Ταυτόχρονα όμως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εάν στηρίξει τις προσπάθειες αυτές, θα μεγαλώσει και την ε, και τον αντίκτυπο των ε, προτάσεων. Τώρα κλείνοντα, θα ήθελα να συγχαρώ την ε, κυρία Μπρέσο και τον κύριο Μπρόκ για τι προσπάθειε που κατέβαλαν στο έγγραφο εργασία για την καλύτερη νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η έκθεσή του τονίζει την ανάγκη τη ε, εμβάθυνση τη ευρωπαϊκή διάσταση δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το μεταναστευτικό, από την οικονομική κρίση, από την κλιματική αλλαγή και τα περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά και την κοινωνική διάσταση και καλωσορίζω επίσης την φιλοδοξία που σας χαρακτηρίζει για να γίνουν αλλαγές στις ε, συνθήκες. Αν και δεν είμαι σίγουρος ε, εάν χρειάζεται αλλαγή συνθήκων για όλες τις προτάσεις που υπάρχουν στην έκθεση. Εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται να εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή όλε τι προτάσει και να αρχίσουμε σήμερα κιόλα για να βρούμε το συντομότερο δυνατόν λύσει έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τι προ... Ε, προκλήσει που υπάρχουν. Όχι μόνο στου τομεί που προανέφερα, αλλά και σε ζητήματα συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια. Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και την καλύτερη εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών και οδηγιών. Τώρα, τα εθνικά κοινοβούλια έχουν ένα όμοιο πρόβλημα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολλές φορές η εκτελεστική εξουσία τους ξεχνά, ιδιαίτερα μάλιστα όταν πρόκειται για ε, διοργανική συνεργασία εκτός ευρωπαϊκών ε, πλαισίων, όπως για παράδειγμα το Fiscal Compact. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ε, πολύ μεγάλη προσοχή ε, σίγουρος ότι το έγγραφο εργασίας ε, θα το συζητήσουμε αργότερα, όμως ήδη μας έχει ζητηθεί να μιλήσουμε για το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Σε σχέση με το σημείο 9 τώρα του εγγράφου εργασίας, που αναφέρεται στη συνθήκη της Λισαβόνας και τα άρθρα 5 και 12, αλλά και το, τα πρωτόκολλα 1 και 2, πιστεύω πως χρειάζεται να γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε αυτά καθώς και στο ρόλο της ε, ΚΟΣΑΚ. Ε, ρητά, ρητή αναφορά. Σχετικά με την διακοινοβουλευτική συνεργασία που αναφέρεται στο σημείο 9 και 10, Αναφέρεται πως δεν θα πρέπει να λαμβάνονται ε, διοργανικές αποφάσεις, αλλά καλύτερα να γίνεται πρώτα μία ανταλλαγή απόψεων όπου τα εθνικά κοινοβούλια θα εξετάζουν αυτά τα ζητήματα και θα υπάρχει μια συντονιστική επίβλεψη έτσι ώστε όλα τα εθνικά κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τα πολύ σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν σήμερα στην ε, συζήτησή μας ε, να είστε σίγουροι πως ε, δεν θα φτάσει ο χρόνος που θα έχουμε. Τα εθνικά κοινοβούλια δεν είχαν εξάλλου πολύ χρόνο, μέχρι 10 μέρες για να, να λύσουν τα έγγραφα εργασίας που τους δόθηκαν. Δεν είχαμε την, την, το χρόνο να το συζητήσουμε ούτε στην Επιτροπή ούτε στις Ολομέλειες. Όμως το non-paper της ΑΦΚΟ σχετικά με την Διοργανική ε, Συμφωνία για καλύτερη νομοθεσία το οποίο, ε, μας, ε, το οποίο μετέφερε η κυρία Χούμπνερ στον πρόεδρο Σούλς έχει μια θετική αντιμετώπιση στην σχέση Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων. Και πιστεύω εδώ πως δεν θα έπρεπε να υπάρχει οποιαδήποτε ανάμειξη που θα επηρεάζει τις αρμοδιότητες και πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει εξηγήσει σχετικά με την επικουρικότητα. Σίγουρα υπάρχουν, πρέπει να υπάρχουν κοινά κριτήρια για την παρατήρηση και τον έλεγχο της επικουρικότητας. Επίσης χρειάζεται και να γίνει μια συζήτηση για το αν ή όχι ε, η διοργανική συμφωνία είναι ο σωστός χώρος για να συζητηθεί η ενίσχυση των ρόλων των ε, κοινοβουλίων. Και τέλος πιστεύω πως μαζί χρειάζεται να συζητήσουμε το πώς θα ενισχύσουμε τον πολιτικό μα διάλογο. Κάτι που θα μπορούσαμε επίση να αναφέρουμε και στο έγγραφο εργασία, διότι η ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου είναι υψή της σημασία για τα εθνικά κοινοβούλια. Στην Βουλή του Λουξεμβούργου Υπάρχει επιθυμία να παίξουμε σημαντικότερο ρόλο στην διαδικασία έγκριση Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και μετά από μια αρχική περίοδο ενθουσιασμού για τη συνθήκη τη Λισαβόνα και εμεί, όπω και άλλα εθνικά κοινοβούλια είχαμε την αίσθηση ότι η, διαδικασία, η επικουρική διαδικασία παρά την ε, μεγάλη τη σημασία. Ίσως ε, δίνει την εντύπωση ότι τα εθνικά κοινοβούλια έχουν περιορισμένο ε, ρόλο και μάλιστα ε, καθυστερούν την ευρωπαϊκή ενοκλήρωση. Χρειάζεται καλύτερα συντονισμένο, περισσότερο πολιτικό διάλογο, ιδιαίτερα στο θέμα της πράσινης κάρτα και πρέπει τα εθνικά κοινοβούλια όντω να παίξουν πιο σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Γι' αυτό λοιπόν θα ε, χαρώ να συνεργαστώ με εσάς, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι αυτό έχει μεγάλη σημασία για, το, ε, για την Βουλή του Λουξεμβούργου και για την Προεδρία μας. Επιθυμούμε μια καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια και αυτό δεν θα γίνει ούτε εδώ ούτε στο Στρασβούργο. Πρέπει να αρχίσουμε από τις πατρίδες μας, καταρχάς σε κομματικό επίπεδο, Δηλαδή, το δικό μου κόμμα, για παράδειγμα, τρεις φορές το χρόνο διοργανώνει συνέδριο με τα μέλη του Κοινοβουλίου. Είναι πολύ σημαντικό μέσα σε ένα κόμμα να μπορούν να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές απόψεων. Από την άλλη, και στις επιτροπές του Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου του Λουξεμβούργου καλούμε τους ε, ευρωβουλευτές της χώρας μας και είναι εύκολο βέβαια ε, να γίνει αυτό, διότι είμαστε πάρα πολύ ε, κοντά στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο, οπότε και οι έξι ευρωβουλευτές μας μπορούν να έρθουν. Είναι λοιπόν κάτι που προσπαθούμε να κάνουμε, μια ανταλλαγή απόψεων σε βάθος και όχι απλά ε, τυπική. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων και σε θεσμικό επίπεδο αλλά και στις πατρίδες μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ Μάρκ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κανονικά ε, ας μην χειροκροτούμε γιατί θα έπρεπε να χειροκροτούμε όλους ε, ομιλητές. Πάμε μέσα στον Υπουργό κύριο Νικολά Σμίτ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί βουλευτές από τα Κοινοβούλια των Κρατών Μελών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ναι, το Λουξεμβούργο είναι υπεύθυνο για την Προεδρία και εγώ είμαι υπεύθυνο για τις σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά οι σκέψεις που θα σας πω είναι πολύ προσωπικές. Δεν θα πρέπει να θεωρήσετε ότι ομιλώ εξ ονόματος επισήμως της Προεδρίας του Συμβουλίου. Αυτά τα οποία θα σας τα πω, θα σας τα πω σαν εκπρόσωπος της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας θέλω και εγώ να συνεισφέρω στην προσπάθεια που κάνετε και είναι μεγάλη η προσωπική μου ικανοποίηση που θα σας μεταφέρω τις απόψεις μου για την θεσμική κατάσταση της Ένωσης και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Κοινοβουλίων των Κρατών Μελών. Διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το έγγραφα εγγρασίας της κυρίας Μπρέσο και του κυρίου Μπρόκ. Πράγματι, καταθέτουν ιδέες χρήσιμες και ενδιαφέρουσες για τη διασφάλιση της συνέχειας της επεξεργασίας των θέσεών μας. Διάβασε επίσης με ενδιαφέρον και την έκθεση Verhofstadt. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μια δημοσκόπηση η οποία έγινε εδώ και λίγες εβδομάδες από το Ίδρυμα Μπέρτελσμαν, το οποίο επισκέφθηκα χτες. Στα αποτελέσματα Τη έρευνα αυτή πρέπει να μας προβληματίσουν. 72% αυτών που να απαντούν, των Ευρωπαίων δηλαδή, των Ευρωπαίων πολιτών, επιβεβαιώνουν ότι η ευρωπαϊκή πολιτική ή οι ευρωπαϊκές πολιτικές αν θέλετε κατευθύνονται προς μια λανθασμένη κατά αυτούς κατεύθυνση. Αυτό επιβεβαιώνει δηλαδή μια ευρωσκεπτιστική τάση στο εσωτερικό των χωρών μας και στο εσωτερικό της Ένωσης μια τάση η οποία φαίνεται ότι είναι αρκετά ισχυρή. Αυτό είναι το κακό κομμάτι, το άσχημο νέο. Υπάρχει όμως και κάτι το θετικό. Το 60% και πάνω από το 60% για τις χώρες της ζώνης ευρώ θεωρούν ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η πολιτική και οικονομική ολοκλήρωση. Νομίζω λοιπόν ότι τίθεται ένα θέμα εδώ για την φύση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Αυτό είναι κανονικό. Στα πλαίσια μιας δημοκρατίας μπορεί κανείς να έχει άποψη για το θετικό ημί των πολιτικών. Αλλά από ό,τι φαίνεται μια ισχυρή πλειοψηφία των Ευρωπαίων <clears throat> θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και από την άλλη βέβαια πιστεύουν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πιο ισχυρή πολιτική και οικονομική ολοκλήρωση. Οι επιθυμίες αυτές των πολιτών για μια ισχυρότερη Ευρώπη, για πιο δραστήρια και ικανή Ευρώπη, που μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις και σήμερα ξέρουμε τι συμβαίνει, βλέπουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, Κάθε εβδομάδα και κάτι συμβαίνει, είτε στον τομέα της μετανάστευσης, της τρομοκρατίας, της ανασφάλειας σε όλα τα επίπεδα. Ας κοιτάξει κανείς τι γίνεται στην ανατολική γειτονία και θα διαπιστώσει τα προβλήματα τα οποία μας περιβάλλουν και τις πραγματικές απειλές. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις στις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών. Να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και γι' αυτό ακριβώς η δική σας πρωτοβουλία είναι μια πολύ θετική πρωτοβουλία συνάντησης με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Δεν χρειάζεται να υπογραμμίσω τη σημασία των κοινοβουλίων μας όχι μόνο για το κάθε κράτος μέλος αλλά και για το σύνολο της Ένωσης. Θυμίζω ότι το άρθρο 12 της συνθήκης προβλέπει ότι τα εθνικά κοινοβούλια συνεισφέρουν ενεργά στη σωστή λειτουργία της Ένωσης και δεν έχουν μια απλή συμβουλευτική περιφερειακή θέση. Αντίθετα κατέχουν μια μίζωνα πολιτική θέση και ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία Έχω την αίσθηση ότι τα κοινοβούλια θα πρέπει να αποκτήσουν ένα ακόμα ισχυρότερο ρόλο. Είναι επίσης προφανές ότι στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, η οποία ελπίζω κάποια στιγμή να οδηγήσει σε μία νέα διακυβερνητική διάσκεψη, ελπίζω λέω, τα, τα κοινοβούλια θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Και όσοι είχαν πάρει μέρος στην προηγούμενη συνέλευση νομίζω ότι θα διαπίστωσαν ότι η συμμετοχή και η συνεισφορά των κοινοβουλίων αυτών στην επιτυχία της συνέλευσης και δεν το λέγω αυτό γιατί είχα πάρει μέρος, ήταν πράγματι επιτυχής αυτή η προσπάθεια. Ο ρόλος των κοινοβουλίων ήταν καθοριστικός. Να μην επανέλθω τώρα στον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι προφανές ότι ο ρόλος αυτός αυξήθηκε, ενισχύθηκε και διευρύνθηκε από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και νομίζω ότι ε, ε, είναι απόλυτα φυσιολογικό πλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι το φόρουμ στο οποίο εκφράζεται η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ε, κρατά ικανοποιημένους. Για την προοπτική αναθεώρηση των συνθήκων. Θα πρέπει να ξεκινήσει κανείς από την υπόθεση ότι η παρούσα διάταξη ε, δίνει την δυνατότητα προσαρμογής, δεν είναι η τελική. Δίνει τη δυνατότητα να επιφέρουμε αλλαγές οι οποίες υπογραμμίζονται από πολλούς και υπογραμμίζονται και στις δύο εκθέσεις ε, της Επιτροπής σας. Όμως θεωρώ ότι υπάρχει ακόμα ένα περιθώριο, υπάρχει ένα ισχυρό περιθώριο. Πρώτον γιατί οι θεσμικές εξελίξεις μπορούν να βελτιωθούν και να επιταχυνθούν σε επίπεδο πρακτικής. Τι εννοώ, η δική σας Επιτροπή αποδεικνύει ε, τον τρόπο εξέλιξης και βελτίωσης των συνεργασιών στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεύτερον, μπορούμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές χωρίς να θίξουμε τη συνθήκη, αλλά βελτιώνοντας τη διαδραστικότητα ανάμεσα στα θεσμικά όργανα. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα και στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης για μια νέα διοργανική. Στόχος της ε, διοργανικής αυτής δεν είναι η τροποποίηση των συνθήκων. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα αυτό. Αλλά στόχος είναι η αναζήτηση του τρόπου με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο μπορούν να δράσουν από κοινού έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια καλύτερη νομοθετική τάξη στην Ευρώπη. Απαιτείται η συνεργασία ανάμεσα στα τρία θεσμικά όργανα, ιδιαίτερα ανάμεσα στα δύο συνομοθετικά όργανα, για να βελτιώσουν τους όρους ακριβώς συνέργειας. Και στη συνέχεια θα δούμε εάν απαιτούνται περαιτέρω ρυθμίσεις σε σχέση με την συνθήκη. Πριν φτάσουμε εκεί και περιλαμβάνεται αυτό στις εκθέσεις, θα πρέπει να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες τις οποίες παρέχει η παρούσα συνθήκη. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες οι οποίες μένει ακόμη να ερευνηθούν. Ας πούμε, στον τομέα της μετανάστευσης. Η αντιμετώπιση της μετανάστευσης δεν είναι κάτι το οποίο, για το οποίο μάλλον δεν μας δίδουν τα μέσα αντιμετώπισης του οι συνθήκες. Τα μέσα υπάρχουν, απαιτείται πολιτική βούληση και απαιτείται μια κοινή πολιτική γραμμή. Και το ίδιο ισχύει επίσης και σε ό,τι έχει σχέση με θέματα ασφαλείας. Νομίζω λοιπόν ότι η συνεργασία με τα κοινοβούλια των κρατών μελών είναι καθοριστική. Μία παρένθεση εδώ. Απαιτείται για όλα αυτά να υπάρξει μία συνοχή στην θεσμική μας αρχιτεκτονική, στην θεσμική μας κατασκευή. Δεν μπορούμε να εμπλέξουμε όπως ζητήθηκε ε, τα κοινοβούλια, τα εθνικά, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής νομοθετικής δραστηριότητας. Νομίζω ότι έτσι και αλλιώς εμπλέκονται τα εθνικά κοινοβούλια και μέσω της διαδικασίας της επικουρικότητας. Εδώ τα εθνικά κοινοβούλια παίζουν ρόλο σημαντικό αλλά δεν μπορούμε να καταστήσουμε τα εθνικά κοινοβούλια έναν τρίτο νομοθέτη στα πλαίσια της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων στην Ένωση. Κάτι τέτοιο ε, θα δημιουργήσει δυσκολίες στο Συμβούλιο καταρχάς. Δεν θα είχε πλέον ρόλο να παίξει το Συμβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι το αίτημα αυτό και γνωρίζετε από πού προέρχεται είναι ένα αίτημα το οποίο είναι ασύμβατο με την θεσμική αρχιτεκτονική την οποία διαθέτουμε. Τελειώνοντας, δύο συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Καταρχάς, η Ευρωζώνη. Εδώ νομίζω ότι απαιτείται στα πλαίσια της ενίσχυσης της Ευρωζώνης να επανεξετάσουμε κάποιες από τις προβλέψεις λειτουργίας. Η διακυβέρνηση της Ευρωζώνης οφείλει να βελτιωθεί και υπάρχουν προτάσεις και μέσω της εκθέσεως των πέντε προέδρων και ε, μέσω της, ε, ε, της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου. Απαιτείται όμως περαιτέρω βελτίωση. Η κατανομή της κυριαρχίας στην Ευρωζώνη θα πρέπει να επιταχυνθεί. Έχω την αίσθηση ότι όλοι βιώσαμε την μεγάλη κρίση, τις απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν, απαντήσεις μερικές φορές ιδιαίτερως βιαστικές και νομίζω ότι απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης. Και θα ήθελα επίσης και για τον δικό μου τομέα, τον κοινωνικό τομέα, να συμπεριλάβουμε τον κοινωνικό τομέα στην διακυβέρνηση της Ευρωζώνης. Εξού και η αναγκαιότητα η εξισορρόπησης ε, της διακυβέρνησης αυτής μέσω και της δημιουργίας φυσικά ενός Eurogroup κοινωνικών θεμάτων. Γι' αυτό δεν απαιτούνται αλλαγέ στι συνθήκε. Μπορούμε να το κάνουμε με πραγματιστικό τρόπο. Και δεύτερον είναι η ενίσχυση η δημοσιονομική της Ευρωζώνης. Και εδώ χρειαζόμαστε κάποιες αλλαγές όμως σε επίπεδο συνθήκης. Γιατί γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια νομισματική ένωση αν δεν υπάρχει μια ισχυρή δημοσιονομική αρμοδιότητα. Και όποιος λέγει δημοσιονομική αρμοδιότητα εννοεί βέβαια ενίσχυση των ιδίων πόρων ακριβώς για τη χρηματοδότηση αυτής της ικανότητας της δημοσιονομικής. Εδώ πρέπει να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις και σε επίπεδο διακυβερνητικών ρυθμίσεων και στο τέλος να αναφέρω το θέμα της δημοκρατικής νομιμότητας. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και σε επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να υπογραμμιστεί και τα κοινοβούλια θα πρέπει να εμπλακούν περισσότερο και σε επίπεδο καθορισμού και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Υπάρχει ένα αίτημα ισχυρό για ένα κοινωνικό πρωτόκολλο, γιατί υπάρχει μια μόνιμη αβεβαιότητα γύρω από τη σχέση ανάμεσα στις τέσσερις ελευθερίες, τις καθοριστικές για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και από την άλλη τις κοινωνικές απαιτήσει και για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και τώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την ιδέα ενός κοινωνικού πυλώνα, θα πρέπει να διευκρινίσουμε τον ρόλο του πυλώνα αυτού σε σχέση με τις τέσσερις ελευθερίες. Δεν θα μπορέσουμε μακροπρόθεσμα να συνεχίσουμε να αφήνουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με όλο το θαυμασμό που του τρέχω φυσικά, την υποχρέωση, γιατί δεν είναι δική του επιλογή, να παίρνει πάντα αποφάσεις ανάμεσα στη μία τις τέσσερις βασικές θεμελιώδεις ελευθερίες και στην άλλη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε επίπεδο απειλών λοιπόν, τις οποίες εφιστάμεθα σήμερα, θα ξεκινούσα λέγοντας ότι κατεπηγόντως πρέπει να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία οι συνθήκες μας επιτρέπουν να εφαρμόσουμε. Η αλληλεγγύη είναι εγγεγραμμένη στη συνθήκη. Υπάρχουν βέβαια κάποια στάδια στα οποία δεν έχουμε ακόμα φτάσει, δεν τα έχουμε ακόμα διανύσει. Σαν παράδειγμα ακούσαμε τι έγινε πρόσφατα με το 47.2, το άρθρο 47.2 ή μάλλον 42.7, συγγνώμη. Νομίζω ότι η αλληλεγγύη θα πρέπει να πάρει μια προφανέστερη μορφή. Δεν μπορεί να υπάρχει μια αλληλεγγύη από τους μεν που διαθέτουν τους σπόρους, που διαθέτουν τις δράσεις, Όταν κάνει κάτι μια χώρα σε στρατιωτικό επίπεδο και το φύγει αυτό οικονομικά, δεν το κάνει μόνο στο όνομά του, δεν το κάνει μόνο για δικούς του λόγους. Το κάνει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα πρέπει να δειχθεί και με την βοήθεια έστω και τη στρατιωτική των υπολείπων χωρών και αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό και μέσω μιας διαφορετικής οικονομικής διαχείρισης. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε μια χώρα ότι δεν σέβεται το σύμφωνο σταθερότητας και ταυτόχρονα η χώρα αυτή να έχει εμπλακεί σε μια τεράστια προσπάθεια διασφάλισης της ασφάλειας σε όλη την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που είπατε και αυτό που επαναφέρατε την πολιτική βούληση που νόμιζα ότι ήταν εκλειπούσα πλέον. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη πολύ στεναρή σας ε, τοποθέτηση και το όραμα ε, και καλύψατε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που μας ενδιαφέρουν και εμά και την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ και τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε τον Διευθύνη κύριο Πασκάλ Ντίνη, προσωπεί τον κύριο Τίμερμαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους σας. Θα ήθελα καταρχάς να σας διαβιβάσω ε, ε, την λύπη και τη συγνώμη του κυρίου Τίμερμανς που κολλείεται σήμερα γιατί τον κάλεσαν επιγόντως εχθές το απόγευμα να πάει στην Τουρκία. Και όπως ξέρετε, είμαστε μέσω διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα δράσης με τις τουρκικές αρχές και χρειάστηκε να επιστρέψει για να συζητήσει κάποια πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία και θέματα αυτού του προγράμματος δράσης. Σήμερα το πρωί θα ήθελα να κάνω μερικά σχόλια για τις σχέσεις μεταξύ της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Εθνικών Κοινοβουλίων. Για να δούμε τι έχει αλλάξει. Βεβαίω για τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων σε εκείνους εναπόκειται να μας πούν αν άλλαξαν κάποια πράγματα, τουλάχιστον εμείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούμε να αλλάξουμε. Πρώτον, όταν ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η νέα, ε, έφερε ένα σύνθημα ότι θα πρέπει να είμαστε μεγάλοι στα μεγάλα πράγματα και μικροί στα μικρά πράγματα. Δηλαδή ε, πώς θα ασχολούμαστε με τις εργασίες μας και πώς θα έχουμε ε, τις σχέσεις μας με ε, τα Εθνικά Κοινοβούλια. Έχουμε ένα πρώτο αντιπρόεδρο που ε, έχει στο χατοφυλάκιό του τα θεσμικά θέματα, ιδιαίτερα τις σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά τώρα έχουμε και μια κοινή ευθύνη και αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ουδέποτε στο παρελθόν είχαν συνεδριάσει τόσο πολλοί επίτροποι ε, ε, με κοινοβούλια, σε επίπεδο κοινοβουλευτικής επιτροπής ή ολομέλειας. Σε ένα χρόνο και κάτι είχαμε πάνω από 200 επισκέψεις σε συνεδριάσεις επιτροπών και ολομελιών σε εθνικά κοινοβούλια, επισκέψεις επιτρόπων. Επίσης, Έχουμε αλληλογραφία, δηλαδή γραπτό διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Από την 1η Σεπτεμβρίου του 2015 έχουμε εισαγάγει ένα νέο τρόπο απάντησης στις αιτιολογημένες νόμες και ε, στις γνώμες που λαμβάνουμε τις νομοδοτήσεις ε, στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και οι απαντήσεις αυτές έχουν μια πολιτική χρειά περισσότερο. Τι συνυπογράφουν ο αρμόδιος επίτροπος εκάστοτε και ο αντιπρόεδρος Τίμερμανς και επισυνάπτουμε στις απαντήσεις τα τεχνικά στοιχεία που λαμβάνουν όλα ε, τα πολιτικά μάλλον όλα τα εθνικά κοινοβούλια μαζί με τις πολιτικές απαντήσεις. Τρίτον, Φέτος το Μάιο εγκρίναμε το πακέτο για την καλύτερη νομοθεσία το ΕΠΝΟΜΟΘΕΤΗΝ, το Better Regulation, που έχει στόχο να εντείνουν και να αυξήσουν τις ε, διαβουλεύσεις και τις ε, συνομιλίες που έχουμε πριν την κατάθεση ε, μιας νομοθετικής πρότασης. Και ενθαρρύνουμε πάρα πολύ τα Εθνικά Κοινοβούλια να αξιοποιήσουν πλήρως αυτή τη δυνατότητα που τους δίδεται πολύ νωρί στο στάδιο μια νομοθετική προπαρασκευαστική διαδικασία να κάνετε προτάσει. Βλέπουμε λοιπόν να μετεξελίσσονται οι σχέσει μα με τα εθνικά κοινοβούλια από τον αριθμό των ε, κυτρίνων ε, καρτών που δραματικά μειώθηκε πέρυσι. Τα τελευταία δύο χρόνια μάλλον είχαμε δύο περιπτώσεις μόνο κίτρινης κάρτας. Ο καθένας μπορεί να ερμηνεύσει με τον τρόπο του αυτή την κατάσταση. Είτε έχει βελτιώσει αισθητά ε, τις δικαιολογήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς την η οτι υπάρχουν άλλοι παράγοντες. Σίγουρα η λήξη της θητείας της προηγούμενης Επιτροπής και η μείωση βέβαια αυτόν τον καιρό των νομοθετικών πρωτοβουλειών εξηγούν από μόνοι τους το γεγονό ότι έχουν μειωθεί και οι κάρτε, αλλά όχι στο βαθμό που εμφανίστηκε. Το ίδιο ισχύει και για την αιτιολογημένη γνώμη. Το ήταν 88, δηλαδή ανησυχίες των Εθνικών Κοινοβουλίων για την επικουρικότητα, πέρυσι 21 και φέτος μέχρι τώρα μόλις 8. Έχω την τάση να πιστεύω λοιπόν ότι είναι θετική αυτή η εξέλιξη, διότι ταυτόχρονα όσο πιο ε, θετική είναι η ατζέντα το θεματολόγιο, Αναπτύσσεται. Πέρυσι είχαμε 600 γραπτές ανταλλαγές απόψεων, αλληλογραφία δηλαδή με τα Εθνικά Κοινοβούλια στον πολιτικό διάλογο με πιο πρόσφατο παράδειγμα ότι για πρώτη φορά στην ιστορία μας είχαμε πράσινη κάρτα, οι συνεισφορέ από 17 κοινοβούλια που προτείνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνουν μια, να κάνουν μια νομοθετική πρόταση για τη σπατάλη των τροφίμων. Ο πρώτο αντιπρόεδρος Τίμερμανς ήδη έχει πει και στην Κόζακ ότι το του αρέσει πάρα πολύ αυτό το σύστημα της πράσινης κάρτας. Εντάσσεται στο πλαίσιο των συνθήκων, δεν χρειάζεται καμία τροποποίηση αν θεώρηση των συνθήκων για να λειτουργεί. Και δύο είναι τα σημαντικά στοιχεία για μας εδώ. Πρώτον, ο χρονισμός, δηλαδή η πράσινη κάρτα από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βουλή των Λόρδων έφτασε ακριβώς την κατάλληλη στιγμή. Διότι προετοίμαζε τότε, εκπονούσε τη νέα νομοθετική δέσμη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κυκλική οικονομία. Δηλαδή δεν μπορούσε να υπάρξει καλύτερη χρονική στιγμή για την κατάθεση αυτή τη πρόταση. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό και επίκαιρο είναι αυτό ο μηχανισμό. Δεύτερον, πολλά κοινοβούλια ή σώματα κοινοβουλίων από το σύνολο των 41 ε, υποστηρίζουν αυτό το μηχανισμό και έχει σημασία αυτό το αριθμητικό στοιχείο γιατί όσο περισσότερα κοινοβουλευτικά σώματα το υποστηρίζουν δείχνουν γνήσιο ενδιαφέρον ε, σε εθνικό επίπεδο και αυτό καταλαβαίνετε ότι αυξάνει το ειδικό βάρος της πρότασης και αναγκάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τη λάβει υπόψη. Και χαίρομαι κύριε Άζελ που αναφερθήκατε στο γεγονός ότι απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την πρώτη πράσινη κάρτα να δούμε πώς θα πάνε οι δύο νέες πρωτοβουλίες. Ελπίζουμε να στεφθούν με επιτυχία. Βεβαίω υπάρχουν και κάποιε λεπτομέρειε που θα πρέπει να συζητήσουν τα εθνικά κοινοβούλια. Ποιο αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία, υπάρχουν όρια για την πράσινη κάρτα. Αν θέλει ένα άλλο εθνικό κοινοβούλιο να προσθέσει, να αφαιρέσει κάτι από την αρχική πρωτοβουλία. Αυτά είναι τεχνικά θέματα και λεπτομέρειες. Πάντως η πρωτοβουλία από μόνη της είναι αξιόλογη. Δεν θα αναφερθώ τώρα σε μια επιστολή που πήραμε την περασμένη εβδομάδα ε, από κάποιο πρωθυπουργό που μίλησε για άλλο μηχανισμό και για κάρτες άλλων χρωμάτων. Καλωσορίζουμε λοιπόν πάρα πολύ και χαιρετίζουμε ε, τη διακοινοβουλευτική συνεργασία και το συντονισμό και πάλι έχει σημασία εδώ ο αριθμός. Δηλαδή, μας χαροποίησε πολύ η πρωτοβουλία που έλαβαν κάποια εθνικά κοινοβούλια να εντοπίσουν στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ποια ε, θέματα θα μπορούσαν να είναι προβληματικά και προσπάθησαν λοιπόν να συνεννοηθούν με ομολόγους τους σε άλλα κράτη-μέλη για να συνεννοηθούν και να φέρουν μια κοινή απάντηση επέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι πάρα πολύ πολύτιμο εργαλείο και εμείς ενθαρρύνουμε και μάλιστα σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο μια τέτοια κοινοβουλευτική συνεργασία και συντονισμό. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση της Ευρωζώνης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, ενέχεται πάρα πολύ ενεργά. Ξέρετε την έκθεση των πέντε προέδρων για την εμβάθυνση της ΟΝΕ, της ε, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Μιλήσαμε για δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση με τις κείμενες συνθήκες, χωρίς τροποποίηση των συνθήκων και σε μια δεύτερη φάση τι θα μπορούσε ρεαλιστικά να ενταχθεί στις συνθήκες. Και είμαστε και φιλόδοξοι για την εξωτερική εκπροσώπηση της Ευρωζώνης και προσβλέπουμε στις συζητήσεις που θα γίνουν εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά και στο Συμβούλιο όπου κάπου, πώς να πω, συνάντησε κάποιες ανησυχίες και προβληματισμούς αυτό. Υποστηρίζουμε λοιπόν στεναρά τη διακοινοβουλευτική συνεργασία και καλωσορίζουμε κάθε πρωτοβουλία ε, ε, στο παρόν πλαίσιο των συνθήκων και ενδεχομένως αν χρειαστούν αλλαγές να σκεφτούμε και αυτές. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία στα σχόλιά σας. Σα ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και όλα τα εθνικά κοινοβουλία. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε τώρα στην ουσία της σημερινής ε, συζήτησης και καταρχάς θα ήθελα να σας ενημερώσω για ένα τεχνικό ζήτημα. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω όσοι έχετε έρθει από τα Εθνικά Κοινοβούλια ότι είστε προσκεκλημένοι για γεύμα στο, ε, στην αίθουσα 4 των ε, μελών. Στο σαλόνι λοιπόν, μετά τις 12.30 δεν ε, θέλω να δεχτώ παράπονα από κανέναν, θα έρθετε. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Περνάμε στην παρουσίαση των δύο εισηγητών της Mercedes Bresso και του Elmar Brock. Ποιος θα πάρει πρώτα το λόγο. Εσείς θα αποφασίσετε. Έχετε όμως 7 λεπτά ο καθένας και σας παρακαλώ να σεβαστείτε το όριο αυτό. Καλημέρα σε όλους. Θα μιλήσω την Ιταλική. Σας καλωσορίζω και εγώ και ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα σας υπενθυμίσω τα φρικτά γεγονότα του Παρισίου, το οποίο προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση και ξέρετε ότι ο πρόεδρος όντως ζήτησε την ενεργοποίηση του άρθρου 42 ζητώντας την αλληλεγγύη και τη στήριξη της Γαλλίας από τις υπόλοιπες χώρες. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και το 222 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ένωσης που προβλέπει την υποχρέωση των κρατών μελών να έρθουν άρρωγοι στην περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης. <clears throat> Το παράδειγμα αυτό νομίζω δείχνει την δυνατότητα που έχει η συνθήκη της Λισαβόνας να δώσει απαντήσεις στις απαιτήσεις για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην Ένωση και σε κοινωνική κατεπίγουσα κατάσταση και σε οικονομική και σε μεταναστευτική και σε πρόβλημα έκτακτο ασφαλείας. Αυτή είναι και η προσπάθεια την οποία κάνουμε στη δική μας έκθεση. Να δείξουμε δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο συμπεριέχει η συνθήκη τα στοιχεία που θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει στον δρόμο ολοκλήρωσης χωρίς να χρειαστεί να περάσουμε με βιαστικό τρόπο σε μεταρρυθμίσεις και σε αλλαγές της συνθήκης. Τα προβλήματα είναι η μεταναστευτική κρίση, η παγκοσμιοποίηση οικονομική, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, οι συνέπειες των κλιματολογικών αλλαγών, οι αδυναμίες της ε, νομισματικής ένωσης στην παγκόσμια κρίση, η έλλειψη ανταγωνιστικότητας, οι κοινωνικές συνέπειες της έλλειψης αυτής, η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και το ψηφιακό πρόβλημα. Να ξεκινήσω από την οικονομική κρίση. <clears throat> Πέρα από την κρίση του δημοσίου χρέους, έδειξαν ότι έχει αδυναμία το σύστημα <clears throat> οικονομικής διακυβέρνησης και αυτό το υπενθύμησε άλλωστε και ο Λουξεμβούργιος Υπουργός. Είναι απαραίτητο να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα μέσα από τα διάφορα πακέτα μέτρων ακριβώς και να εξυπηρετήσουμε τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και των πολιτών και να καταστήσουμε τις διαδικασίες τις οποίες ακολουθούμε και στον οικονομικό τομέα πιο δημοκρατικές και διαφανείς. Και θα πρέπει επίσης να ενισχύσουμε και τον μηχανισμό σταθερότητας. Για να το πετύχουμε αυτό απαιτείται μια περαιτέρω ολοκλήρωση της Ευρωζώνης η οποία στην ουσία απαιτεί να υπάρξει ένας προϋπολογισμός ισχυρότερος της Ευρωζώνης που θα επηρεάζει τις οικονομικές εξελίξεις και θα αποτρέπει τις κρίσεις. Η ενιαία αγορά, η μεγαλύτερη κατάκτηση της Ένωσης θα συντηρηθεί σωστά και όπως είπατε άλλωστε υπάρχει η δυνατότητα στο εσωτερικό της συνθήκης λήψης υπόψη και της κοινωνικής διάστασης. Δεν είναι μόνο οικονομικό πρόγραμμα αλλά είναι και κοινωνικό και απαιτείται βέβαια η οικονομική ανάπτυξη, αλλά για κοινωνικούς λόγους. Πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν την κοινωνική αυτή διάσταση, πρέπει να εγγυηθούμε καλύτερα τα δικαιώματα των κινητικών σε εισαγωγικά εργαζομένων και να διασφαλίσουμε και τα κοινωνικά δικαιώματα όπως θα προβλέψουν τα άρθρα 151 και 153. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε επίσης την ιδέα ενός ελαχίστου μισθού που θα αποφασίζεται από τα κράτη-μέλη σε σχέση με τα επίπεδα εισόδων. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι η εξωτερική διάσταση και η ασφάλεια και η άμυνα. Οι λόγοι είναι προφανείς. Νομίζω ότι αναπτύσσοντας μια κοινή εξωτερική πολιτική στον τομέα αυτό θα έχουμε βασικά πλεονεκτήματα θα αντιμετωπίσουμε την αναποτελεσματικότητα των πολλαπλών φωνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα έξω, έχει φτάσει η στιγμή να αναγνωρίσουμε ότι μόνο σαν Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις. Υπάρχει λοιπόν μια ολόκληρη σειρά προτάσεων, όπως η μετατροπή του Frontex σε Ευρωπαϊκή Σύνοριοφυλακή και διαφορετικές μορφές συνεργασίας για την φύλαξη των συνόρων της Ένωσης είναι κάτι το απαραίτητο. Ε, η θεσμική οργάνωση τώρα, δεν έχω να μιλήσω για αυτό χρόνο όσο θα ήθελα. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών Θα πρέπει το Συμβούλιο στο εσωτερικό της συνθήκης να μπορέσει να λειτουργήσει σαν νομοθετικό σώμα, έτσι ώστε οι υπόλοιποι κοινοτικοί σχηματισμοί να λειτουργούν σε προπαρασκευαστικό επίπεδο. Θα πρέπει να καθοριστούν επίσης και οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που τα τελευταία χρόνια θα έλεγα έχει λίγο ξεχυλήσει προς διάφορες κατευθύνσεις. Θα πρέπει επίσης έστω και επιμέρους να υπάρξει μια αντιμετώπιση του ρόλου των κοινοβουλίων των κρατών μελών. Η στιγμή η τωρινή είναι μια καλή στιγμή για να προτείνουμε τροποποιήσεις, αλλά νομίζω ότι η συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών θα πρέπει να ενισχυθεί. Ας ελέγξουμε πώς θα λειτουργήσει ή πώς δεν έχουν λειτουργήσει μέχρι τώρα οι κίτρινες και πορτοκαλί κάρτες. Θα πρέπει να δούμε επίσης και τι συμβαίνει ε, μετά από την επιστολή του Πρωθυπουργού Κάμερον και να δούμε τι είδους διαπραγματεύσεις θα έχουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο. Νομίζω ότι η πράσινη κάρτα θα μπορούσε να λειτουργήσει ορθότερα και επί τη βάση και των σημερινών συζητήσεων θα μπορούσαμε να σκεφτούμε πώς μπορεί να διαρθρωθεί η διαδικασία αυτή της πράσινης κάρτας με διαδικασίες διαφανέστερες και ευκρινέστερες. Λοιπόν, τελειώνω. Μου λέγουν ότι δεν έχω άλλο χρόνο στη διάθεσή μου. Νομίζω λοιπόν ότι ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η διαδικασία λήψεως αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το θέμα της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία ή ενισχυμένη πλειοψηφία ή και ομοφωνία. Αυτά είναι θέματα που μας απασχολούν στη δική μας έκθεση, γιατί νομίζουμε πράγματι ότι έχει μεγάλη σημασία να χρησιμοποιήσουμε και την ειδική πλειοψηφία περισσότερο από την, από την ομοφωνία και υπάρχει πάντα περισσότερη χρήση τη διαδικασία ενισχυμένη συνεργασία ανάμεσα σε συγκεκριμένα κρατημέλη. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Σαν εισηγητές εμείς περιμένουμε με ενδιαφέρον τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ελμαρμπρόκ θα πάρει το λόγο. Σας θυμίζω, ε, αν θέλετε να μιλήσετε, να μας ε, το δηλώσετε το συντομότερο για να δούμε πώς θα μοιράσουμε το χρόνο. Ο Έλμαρ Μπρόκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Η κυρία Μπρέσο και εγώ πονήσαμε ένα σχέδιο έκθεσης και εν ώψη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε ως Ευρωπαίοι σε αυτή την παγκόσμια τάξη. Πιστεύω ότι ο τρόπος εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρμοδιότητες της θα πρέπει να προσανατολίζεται ε, στο εξή, με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίζουμε καλύτερα τις προκλήσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και η συνθήκη της Λισαβόνας δίδει πολλές δυνατότητες που ακόμα δεν έχουν αξιοποιηθεί. Αυτό είναι προφανές. Η κυρία Μπρέσο έδωσε μια σειρά από παραδείγματα. Πάντα μας εκπλήσουν, μας ευνηδιάζουν διάφορες κρίσεις τις οποίες δεν είχαμε προετοιμαστεί διότι αποφύγαμε να αξιοποιήσουμε νωρίτερα και προληπτικά δυνατότητες που μας δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας για να έχουμε δημιουργήσει εκείνη την αρχιτεκτονική και τα μέσα για να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις. Αυτό έγινε και με την χρηματοπιστωτική κρίση το 2008 Εάν είχαμε τότε την θεσμική αρχιτεκτονική που με τόσο κόπο χτίσαμε τα τελευταία πέντε χρόνια, τότε θα μπορούσαμε να έχουμε αποτρέψει την κρίση ή να μας είχε βγει πιο φτηνή, εν πάση περιπτώσει. Για τα θέματα τα μεταναστευτικά βρισκόμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Είμαστε τελείως αβοήθητοι, ανήμποροι παρόλο που υπάρχει η δυνατότητα και περιγράφεται ε, πώς φυλάζει κανείς τα εξωτερικά σύνορα. Και η ίδια μου η χώρα πριν από 11 χρόνια αρνήθηκε να χαρακτηρίσει ασφαλείς χώρες ε, τις Βαλκανικές. Ή πριν από 5 χρόνια που είχαμε ε, προβλήματα στη Λαμπεντούσα, αρνήθηκαν τις ποσοστώσεις. Και ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι έρχονται πρόσφυγες και στη Γερμανία και κάποιοι που ήταν κατά των ποσοστώσεων ξαφνικά είναι υποστηρικτές και βγαίνουμε και εκπλησόμαστε γιατί οι άλλοι δεν έχουν κάνει αυτή τη στροφή. Όλα αυτά απερίφθησαν παρόλο που δίνουν οι συνθήκες τη δυνατότητα. Παρίσι, Λονδίνο, Βερολίνο και Άμστερνταμ και από όλη την Ευρώπη ε, βγαίνουν και δηλώνουν ότι υπάρχει πρόβλημα με τις αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υβρίζουν την Ευρώπη που δεν τα έκανε όλα αυτά νωρίτερα ότι απέτυχε πάλι και η Ευρώπη που δεν είναι αλληλέγγυα και πάει λέγοντας. Ε, το επόμενο θέμα. Από την Τρίτη βλέπουμε στον τύπο ότι ο πρόεδρος Ολάουντ ζητεί να κινητοποιηθεί, να ενεργοποιηθεί το άρθρο 42 42-7 της συνθήκης. Και ουδής γνωρίζει τι θα το κάνει αυτό και τι σημαίνει. Η συνθήκη της Λισαβόνας όμως, εξ όσο γνωρίζω, ισχύει εδώ και πέντε χρόνια. Ποιος έβγαλε συμπεράσματα για να έχουμε μια κοινή δράση, ένα κοινό στρατηγείο για να κάνουμε σχεδιασμό, πώς θα γίνει ο επιμερισμός της εργασίας και τι θα κάνουν τα κράτη-μέλη, πώς θα συνεργάζονται, όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μεταξύ τους. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, από πω τι κακό μας βρήκε. Αυτό διαπιστώνουμε ή η μόνιμη διαρθωμένη συνεργασία ως εργαλείο για να μπορούν οι χώρες που το επιθυμούν σε τέτοιες κρίσεις να έχουν ισχυμένη συνεργασία και όσοι δεν το θέλουν να μείνουν απ' έξω. Το λέει η συνθήκη αυτό, υπάρχει δυνατότητα ε, διαφορετικών συμμαχιών κάθε φορά και συνεργασιών. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, ας πούμε, ότι ορισμένε χώρες μέλη δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Όλα αυτά προβλέπονται στη συνθήκη της Λισαβόνας. Εμείς τι κάναμε μέχρι τώρα, τίποτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανούμε 190 δισεκατομμύρια ευρώ, ε, τα κράτη-μέλη δηλαδή για την άμυνα, περισσότερο από τη Ρωσία και έχουμε διπλάσιο στρατό από τους Αμερικανούς, αλλά δυστυχώς δεν ε, έχουμε ενιαία όπλα. Έχουμε 80% ε, αύξηση του κόστου στο στρατό μας, ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλά δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε γιατί δεν έχουμε λέει τι αρμοδιότητε. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα που προβλέπει η συνθήκη και με τρόπο ε, πιο έντονο. Η συνθήκη αυτή έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη. Γνωρίζει ο καθένα από εμά ότι δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει μόνο του αυτά τα ζητήματα. Το μεταναστευτικό, το θέμα της εξωτερικής πολιτικής, της αμυντικής, καταπολέμηση τρομοκρατία, καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής και συνεχίζεται ο κατάλογος. Καμία χώρα δεν μπορεί από μόνη της να τα λύσει αυτά. Καμία. Και κανένα από τα ερωτήματα. Θα πρέπει λοιπόν να καθίσουμε να σκεφτούμε το όποιο στενό, δεν λέω πλαίσιο της συνθήκης που έχουν κυρώσει όλα τα κράτη-μέλη, να βρούμε μια απάντηση. Να προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Και αυτό είναι θέμα της πολιτικής τάξης. Και στα Εθνικά Κοινοβούλια, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν το νοιάζει το πολίτη ποιος είναι ο αρμόδιος ε, θεσμικά. Αδιαφορεί, ούτε αλλάζουν οι αρμοδιότητες. Γι' αυτό η κυρία Μπρέσο και εγώ δεν μιλούμε καθόλου για αναθεώρηση των συνθήκων. Με κείμενε συνθήκε τι μπορούμε να κάνουμε, που μπορούμε. Έχω πλήρη επίγνωση ότι όπω έχει σήμερα το πολιτικό στερέωμα και η ε, ατμόσφαιρα και το κλίμα δεν μπορεί να επιβληθεί η λογική αναθεώρηση των συνθήκων. Ερωτώ λοιπόν αυτά τα προβλήματα πώς μπορούν να λυθούν και κάποια άλλα ακόμα με κοινή πολιτική. Απάντηση. έχουμε θα πρέπει να διαφυλάξουμε πρώτα απ' όλα την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είδαμε και στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο και αλλού. Όλα τα κράτη-μέλη δέχτηκαν ότι το ευρώ είναι το νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία χώρα έχει opt-out και μια άλλη χώρα έχει opt-in. Όλες οι υπόλοιπες υπόκεινται σε κανόνες. Και τώρα να δημιουργούμε νέα θεσμικά εμπόδια ή να έρθουμε να αρνηθούμε ότι είναι το νόμισμά μας το ευρώ. Και όταν έχεις opt-out δεν μπορείς να βγαίνεις και να δικαιολογείς να υπάρχουν διαφορετικά νομίσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά νομίσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το νόμισμα της Ένωσης είναι το ευρώ. Και δεν θέλω τώρα να διχαστούν θεσμικά οι χώρες, σε χώρε του ευρώ και χώρε εκτός ευρώ, σε χώρε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Δεν επιτρέπονται τέτοια πράγματα. Και επίσης αυτό το πλαίσιο κάναμε στην έκθεσή μα πρόταση για τη μετεξέλιξη της ε, ΟΝΕ, πώς μπορούν περισσότερο να συμμετέχουν τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό. Και όσο προχωράει και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε και αυτό είναι ζήτημα αρχής, ότι οι εκάστοτε κοινοβουλευτικές αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται στο εκάστοτε αρμόδιο επίπεδο και ποτέ να μην υπάρχει ανάμειξη γιατί δεν πρόκειται να λειτουργήσει ούτε να έχει ποτέ τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Γι' αυτό αυτό ε, στο μηχανισμό σταθερότητα, στον ESM που τα κονδύλια αυτά ε, είναι των κρατών μελών, η αρμοδιότητα παραμένει στα εθνικά κοινοβούλια και δεν είναι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εάν ήταν σε επίπεδο αλλαγής ε, για τη σύγκληση και άλλα θέματα νομοθεσίας, τότε θα ήταν αρμόδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, θα πρέπει να δούμε ότι, για να καταλάβουμε, πώς θα συνεργαστούμε κοινοβουλευτικά. Στη μετεξέλιξη ή στην υλοποίηση της ειδήξης Λισαβόνας θα πρέπει να φροντίσουμε από κοινού να είναι πιο σαφείς οι δομές λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θέλω να τονίσω κάτι που είπε η στην υλοποιηση της ειδικης λισαβονας θα πρεπει να Μπρέσο. Επιτέλους χρειαζόμαστε ειπε η κυρια μπρεσο τελος χρειαζομαστε διαφανεια στο Συμβούλιο. Έχουμε την κλασική μορφή ε, δύο σωμάτων. Συμβούλιο, Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο όμω δεν λειτουργεί. Μιλώ πάντα για το νομοθετικό επίπεδο. Σαν να έχουμε δύο σώματα. Η κοινοβουλευτική διάσταση του Συμβουλίου δεν λειτουργεί σωστά όπω θα ήταν ένα δεύτερο σώμα κοινοβουλευτικό. Πρέπει και μπορεί να αλλάξει ο κανονισμό του Συμβουλίου. Το έχουμε συζητήσει αυτό και με του πολίτε. Ότι λόγω αυτή τη μεθόδου που ακολουθεί το Συμβούλιο δεν γνωρίζει ο πολίτη Ποιο είναι αρμόδιο και υπεύθυνο για ποια απόφαση. Οι κυβερνήσει κρύβονται πίσω από αυτό και δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για τι αποφάσει που παίρνουν στο Συμβούλιο, απέναντι σε Εθνικά Κοινοβούλια και απέναντι στην κοινή γνώμη. Γι' αυτό θα πρέπει εμεί να δημιουργήσουμε αυτή τη διαφάνεια, να νομοθετεί δημοσίω ε, το Υπουργικό Συμβούλιο και να προετοιμάζουν τις αποφάσεις του Συμβουλίου τα επιμέρους Συμβούλια Υπουργών. και να λαμβάνονται λήψεις κατά πλειοψηφία, ε, να λαμβάνονται συγγνώμη αποφάσεις κατά πλειοψηφία. Τώρα στο Συμβούλιο αυτό δεν συμβαίνει. Και βγαίνουν οι υπουργοί και λένε Μα το γράφει η συνθήκη της Λισαβόνας αλλά δεν το χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι ολέθριο για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και για τους πολίτες. Αφού το λέει η συνθήκη. για σκεφτούμε πώ μπορεί κανεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μπορεί να προσφύγει κατά του Συμβουλίου γιατί είναι μια διαρκή και μόνιμη παραβίαση τη συνθήκη. μπλοκάρουν τα διάφορα θέματα, τι διάφορε αποφάσει και αυτό ε, μα βγαίνει όλο και πιο ακριβό τελικά. Εμεί, ω Κοινοβούλιο θα πρέπει να μπορούμε να το ελέγχουμε και εμεί στο δικό μα επίπεδο και εσεί στο δικό σα επίπεδο και να ενισχυθεί ο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Γι' αυτό τα όργανα που δημιουργήθηκαν για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, ε, το άρθρο 13 και άλλα, για μένα είναι σωστά. Αλλά πάντα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα όργανα δεν είναι όργανα λήψης αποφάσεων. Είναι ε, διαβούλευσης, πληροφόρησης, ενημέρωσης και εκεί υπάρχει συνένεση. Ε, προσωπικά ήμουν αρμόδιος για την ΚΕΠΑ και την ΕΠΑ, Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, και σκέφτομαι την τελευταία συνεδρίαση που είχαμε στο Λουξεμβούργο υπό Λουξεμβουργενή Προεδρία. Και τώρα που υπάρχει η συμφωνία για το άρθρο, 13, άρθρο 13 για την ΟΝΕ, και αυτό ισχύει για το Κοινοβούλιο, για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Ήταν πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμπεριλαμβάνονται και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ε, κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να γίνει και σε αυτό το τομέα. Θα πρέπει να ενημερωνόμαστε, να συζητούμε, να ανταλλάσσουμε πληροφορίε τα Εθνικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ασκούμε ε, τι αρμοδιότητε που έχουμε και να μπορούμε να ελέγχουμε κοινοβουλευτικά ο καθένα στο επίπεδό του. Αλλά να γίνεται σωστά ο διάλογο για να μην διαλυθεί ο κοινοβουλευτισμό πορτοκαλί κάρτες. Τι λέει η συνθήκη. Εάν 50% των κρατών μελών, των εθνικών κοινοβουλίων δηλαδή, διορθώνει ο κ. για λόγους αλληλεγγύη, ε, επικουρικότητας και αναλογικότητας, τις δύο αρχές αυτές, επικουρικότητας και αναλογικότητας, θεωρούν ότι η νομοθετική πρόταση είναι λανθασμένη, τότε εθνικά κοινοβούλια είτε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίς να έχει λόγο Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να τερματίσουν την νομοθεσία. Αυτό εξ όσων γνωρίζω δεν έχει αξιοποιηθεί ούτε μία φορά από κανένα εθνικό κοινοβούλιο. Στην πράξη μπορούμε να συζητούμε ό,τι θέλετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δίνει μεγαλύτερε προθεσμίε πριν την αρχή των 8 εβδομάδων τεχνικά και γλωσσικά. Μπορούμε να βοηθήσουμε και εμεί το Κοινοβούλιο και στη συνεργασία καλύτερα των Εθνικών Κοινοβουλίων, καμία αντίρρηση. Και μπορώ να σας πω ότι και αν το Συμβούλιο στις διαπραγματεύσεις βγαίνει και λέει ότι αν 55% των Εθνικών Κοινοβουλίων και ε, υπάρχει και πλειοψηφία στο Συμβούλιο, ε, είμαστε υποχρεωμένοι, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να τερματίζει τη διαδικασία αυτή τη νομοθετική το Συμβούλιο. Όλα αυτά τα λέει η συνθήκη της Αβώνας. Άλλε συμφωνίες ε, πέρα και έξω από τις ειδήξει τη αγώνα θα είναι πολύ δύσκολες. Γι' αυτό ε, μιλώ για την ενισχυμένη συνεργασία των κοινοβουλίων ε, για να εξασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή τη συνθήκη. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλμαρ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, η οποία ετοίμασε μια γνωμοδότηση και θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να μείνετε εντό του ορίου των 5 λεπτών. Δίνω το λόγο τώρα στον Κονσάλο Λόμπο Ξαβιέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω πως ε, συμφωνούμε και εμεί σε γενικέ γραμμές με τις παρεμβάσεις που ακούσαμε μέχρι τώρα και θα ήθελα να τονίσω και κάποια άλλα σημεία από πλευρά τη δική μα επιτροπή ε, που ε, αφορούν την οργάνωση τη κοινωνία των πολιτών. Ε, Δίχω αμφιβολία, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τι τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην ιστορία της. Όχι μόνο την οικονομική και κοινωνική κρίση που έχει κατακαιρματίσει την κοινωνία μας και έχει δημιουργήσει χάσματα ανάμεσα σε ανθρώπους, σε περιφέρειες και χώρες, αλλά και όπως ακούσαμε σήμερα η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια πάρα πολύ σοβαρή εξωτερική απειλή και απειλή στην ασφάλειά της που απειλεί την Ευρωπαϊκή Συνοχή και Αλληλεγγύη. Και υπό αυτό το πλαίσιο λοιπόν οι ευρωπαϊκές συνθήκες παρέχουν ανεκμετάλλευτες μέχρι τώρα ευκαιρίες για διάφορες πολιτικές και διάφορες διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν και να ενισχύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Η δική μας Επιτροπή θεωρεί ότι αν και στο μέλλον θα είναι αναγκαίο να γίνει μια αναθεώρηση ορισμένων στοιχείων των συνθήκων, ίσως μέσω αλλαγών των συνθήκων, οι προϋποθέσεις για να γίνει αυτό δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν γίνεται να επαναδιαπραγματευτούμε τις συνθήκες αυτή τη στιγμή, διότι έτσι θα ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας. Δεν υπάρχει ούτε πολιτική ούτε και διοικητική βούληση για να γίνει κάτι τέτοιο. Η γνωμοδότησή μας αναφέρεται στο τι μπορεί να γίνει υπό τις παρούσες συνθήκες. Υπάρχουν προτάσεις για την ε, χρησιμοποίηση των, πέτη, των ε, 5 ε, ρητρών από τα άρθρα 5 έως 8. Αυτές οι ρήτρες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να προωθήσουν την ε, διασύνδεση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές ε, πολιτικές και την κινητικότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Επίσης, σε σχέση με την Ενεργειακή Ένωση και την εσωτερική αγορά, υπάρχει η χάρτα των ε, θεμελιωθών ε, δικαιωμάτων, υπάρχει μακροπεριφερειακή στρατηγική για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει και μια επιτακτική ανάγκη μεταρρύθμισης του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η Ευρωπαϊκή και Νομισματική Ένωση χρειάζεται επανέξεταση. Εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ολοκλήρωση μέσω του ε, μηχανισμού της ε, Νομισματικής Ένωσης που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όχι μόνο οικονομικό πυλώνα αλλά και έναν πυλώνα κοινωνικό. Και να σας υπενθυμίσω ότι στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υπάρχει μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλία σχετικά με αυτό το συγκεκριμένο θέμα συμπληρώνοντας δηλαδή τον πολιτικό και οικονομικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι στη γνωμοδότησή μας ε, έχουμε επικεντρωθεί περισσότερο στην αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών της ε, συμμετοχικής ε, δημοκρατίας, της συμμετοχικής διακυβέρνησης, της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Όχι μόνο επιχειρηματολογούμε υπέρ της επιτυχούς εφαρμογής του άρθρου 11 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ζητούμε μια επιστροφή στις παραδοσιακές αξίες, σε ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα στην οικονομική διακυβέρνηση και επίσης είμαστε υπέρ στην ενίσχυση της επικουρικότητας, τόσο οριζόντια όσο και κάθετα με μεγαλύτερες εξουσίες για τους κοινωνικούς εταίρους, για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Και στο πλαίσιο αυτά Ζητούμε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρηση των συνθήκων να συμπεριλάβει την αναγνώριση του ρόλου της Ευρωπαϊκής και Κοινωνικής Επιτροπής στην εφαρμογή του άρθρου 11 της ε, συνθήκης και ζητούμε επίσης να αναγνωριστεί ε, ρητά ο θεσμικός ε, της ρόλος στα πλαίσια της προσπάθειας για καλύτερη νομοθεσία. Σίγουρα δεν είναι εύκολο θέμα αυτό, όμως Δεδομένης της τόσο μεγάλη αστάθεια που υπάρχει τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της Ένωσης, η Επιτροπή μας είναι πεπισμένη ότι μόνο με την περισσότερη ολοκλήρωση θα γίνει πιο ισχυρή η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι χτίζοντα τύχη ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ε, θέτει η γνωμοδότησή μας λοιπόν το, την προσοχή τη στο όραμα για το μέλλον. Κανείς όμως, ούτε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ούτε η κοινωνία των πολιτών, ούτε τα κράτη-μέλη δεν μπορούν μόνα τους να ε, φέρουν εις πέρα σε αυτήν την αλλαγή. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε αλλά να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό που μας δίνει η συνεργασία. Σας ευχαριστώ και ευχαριστούμε την Επιτροπή σας για την προετοιμασία της νομοδότησης και για το σεβασμό του χρόνου από πλευρά σας. Θα δώσω το λόγο τώρα σε όλους τους εκπροσώπους των κοινοβουλίων των κρατών μελών αλλά και των συναδέλφων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λόρδος Μπόσουελ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ εσάς και την Επιτροπή σας για την οργάνωση αυτής της σημαντικής συνάντησης για τις μελλοντικές θεσμικές εξελίξεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η διακοινοβουλευτική συνάντηση έχει σαν στόχο την βελτίωση του πολιτικού διαλόγου ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Έρχεται σε πολύ εύθετη χρονική στιγμή. Εφόσον αποφασίσει να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Κάτω Βουλή αλλά και οι περιφερειακές συνελεύσεις θα θέλουν να συνεργαστούν μαζί σας ακόμα περισσότερο. Οι σχέσεις ανάμεσα στα κοινοβούλια από τη μία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την άλλη δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται από εμπόδια τα οποία δεν χρειάζεται να υπάρχουν. Σας είχα στείλει μια επιστολή για ένα τέτοιο εμπόδιο και εξέφραζα τις ανησυχίες μου. Και νομίζω όπως είπατε ότι συμφωνείτε μαζί μου και το θέσατε και εσείς το θέμα. Στόχος λοιπόν της παρέμβασής μου σήμερα είναι να εξηγήσω ότι η ρύθμιση των δράσεων ε, της, ε, των κρατών μελών, των κοινοβουλίων των κρατών μελών, δημιουργεί δυσκολίες με τον ασυντόνιστο τρόπο που γίνεται στο Westminster. Αυτές οι δυσκολίες έχουν συνέπειες στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους νομοθέτες, τους συνομοθέτες για τον κανονισμό Europol, αλλά και για την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το δικαίωμα έρευνας. Και στα πλαίσια επίσης και του νέου κανονισμού Eurojust θα συμβεί το ίδιο. Ε, το κείμενο εργασίας της ΑΦΚΟ σχετικά με τη βελτίωση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των δυνατοτήτων που δίδει η ε, συνθήκη. Στις παραγράφους 9 και 10 στην ουσία λέγεται ζητείτε prescription των δράσεων των κοινοβουλίων αυτών. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν κοινά σώματα κοινοβουλευτικά τα οποία θα παίρνουν αποφάσεις. Να σας εκφράσω πιο συγκεκριμένα τις ανησυχίες μου εδώ. Σύμφωνα με το Βρετανικό Σύνταγμα, κάποια θέματα δεν διευκρινίζονται κατά λέξη, αλλά είναι σαφές ότι η κάτω βουλή είναι κυρίαρχη μπορεί να προωθεί νομοθετικές ρυθμίσεις και να μην ελέγχεται από τα δικαστήρια. Αυτή είναι βασική αρχή της συνταγματικής τάξης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν μπορεί λοιπόν το Westminster, η κάτω βουλή, να υπόκειται στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που εμπλέκεται σε όσο ναι. κοινοβουλευτικός έλεγχος των εξωτερικών υπηρεσιών. Αυτά περιλαμβάνονται και στην συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι δηλωτικά των ρόλων των κοινοβουλίων των κρατών μελών, στα οποία δεν αποδίδουν συγκεκριμένες νομικές ευθύνες. Το 4.2 επιβάλλει καθήκον στην Ευρωπαϊκή Ένωση να σέβεται τις συνταγματικές δομές των κρατών μελών. Οι δυσκολίες τις οποίες έχω εγώ σε σχέση με το Westminster ίσως να τις έχουν και άλλα κοινοβούλια και θα ήθελα να μάθω ποιες είναι οι απόψεις των άλλων χωρών. Θα ήθελα όμως να τονίσω, Πρόεδρε, ότι οι ανησυχίες μας περιορίζονται στο επίπεδο της διαδικασίας, μέσω του οποίου θα συμφωνηθεί η έρευνα, η διακοινοβουλευτική ή κοινοβουλευτική όπου προβλέπεται. Όχι με την ουσία. Επί της ουσίας εμείς θέλουμε να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια, ε, παραπέμποντας ε, όχι βέβαια απλά στην αναφορά της συνεργασίας αυτής και να μην αφήνουμε τις λεπτομέρειες της συνεργασίας να αποφασίζονται από αυτούς οι οποίοι είναι εκτός θεσμικών οργάνων. Μέχρι τώρα δυστυχώς αυτή ήταν η λογική. Επιτρέπει μένα την διακοινοβουλευτική συνεργασία να αποφασίζεται με συνένεση από τα κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι από τους συνομοθέτες κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων από τις οποίες αποκλείονται τα εθνικά κοινοβούλια. Θέλουμε εμείς μια καλύτερη βάση για αυτή τη μορφή συνεργασίας. Η Άνω Βουλή, όπως ξέρετε, είναι υπέρ της στενότερης συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι μια αναπόφευκτη σύγκρουση για το διαδικαστικό κομμάτι της κοινοβουλευτικής συνεργασίας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφευθεί στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως πάντα μιλάω Ολλανδικά και ε, επειδή υπάρχει και Ολλανδική καμπίνα για να σεβόμαστε και την Ολλανδική γλώσσα. Πρόεδρε, χαίρομαι που βρισκόμαστε εδώ και εγώ αισθάνομαι εσά στο σπίτι μου ε, ως πρώην Ευρωβουλευτής, αλλά θα μιλήσω εξ ονόματος της Ολλανδικής Γερουσίας. Κοιτάξτε, ε, τα προβλήματα που έχουμε σήμερα ποια είναι. Προσωπικά, εδώ και χρόνια εγώ υποστηρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ήμουν μέλος 25 χρόνια θα πρέπει να συνεργάζεται με τα Εθνικά Κοινοβούλια και θα πρέπει ο ένας να είναι το μακρύ χέρι του άλλου στον έλεγχο της γραφειοκρατίας, στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Άρα τι σημαίνει αυτό Πρόεδρε, ότι τα κοινοβούλια θα πρέπει να συνεργάζονται καλύτερα και περισσότερο μεταξύ τους. Κοίταξα και μελέτησα πάρα πολύ το κείμενο που μας δώσατε, αυτό το έγγραφο εργασίας. Και τι βλέπω εκεί. Πολλές προτάσεις βελτίωσης για το... και πώς αυτές μπορεί να γίνουν με τις κείμενες συνθήκες, χωρίς καμία τροποποίηση. Χαίρομαι λοιπόν, Πρόεδρε, που ε, ζητείτε να δοθεί περισσότερη προσοχή στη βελτίωση του εργαλείου που λέγεται κίτρινη κάρτα. Αυτό που διαπιστώνω τώρα, τουλάχιστον στην Ολλανδική Βουλή, είναι ότι υπάρχει μια δυσφορία με το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Και σας παραπέμπω ε, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ένα μόνο παράδειγμα. Ωραία λοιπόν η βελτίωση, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται, και το λέει αυτό το έγγραφο εργασίας, μεγαλύτερη διαφάνεια στο Συμβούλιο την νομοθετική του διάσταση και διαδικασία. Αυτό ισχύει οπωσδήποτε και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω όμως την εμπειρία μου και ως Ευρωβουλευτής 25 χρόνια ότι όταν εδώ ολεκριώνεται σε πρώτη ανάγνωση μία νομοθεσία υπάρχει δυνατότητα ε, δράσεις, ε, η οποία όμως από εκεί πέρα περιορίζεται και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να γίνουν διαφορετικές συνεννοήσεις εκεί και συμφωνίες. Δηλαδή, περισσότερο να εργαζόμαστε, περισσότερες κίτρινες κάρτες, καλύτερες συμφωνίες για την νομοθετική διαδικασία. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν χωρίς να αλλάξουν σημαντικά οι συνθήκες. Αυτό που με προβληματίζει είναι το εξής. Η Προεδρία του Συμβουλίου και η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, ότι πρέπει να συνεργάζονται. Αυτό μπορεί να γίνει χωρίς ε, τροποποίηση των συνθήκων. Εγώ νομίζω όχι. Άρα όσοι κάνουν μια τέτοια πρόταση θα πρέπει να μου πούν πώς γίνεται αυτό χωρίς να αλλάξουν οι συνθήκες. Κάτι άλλο που μου αρέσει πολύ επίσης είναι ότι και θεσμοί όπως η ΟΚΕ αλλά και η Επιτροπή Περιφερειών αναφέρονται στο έγγραφο. Πριν εκλεγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήμουνα και ε, βουλευτής στην Ολλανδία. Δηλαδή έχω εξαντλήσει περίπου το φάσμα. Βουλευτής, ευρωβουλευτής και τώρα είμαι στη Γερουσία. Ε, στη Βουλή όμως ε, των κάτω χωρών ισχύει αυτό, ίσως και σε άλλες χώρες, δεν ε, αποφασίζεται καμιά νομοθεσία χωρίς να έχουν γνωμοδοτήσει οι αρμόδιες επιτροπές, η ΟΚΕ δηλαδή, η Επιτροπή Περιφερειών, η αντίστοιχη της χώρας μου. Εναπόκειται όμως στις δύο αυτές επιτροπές, οικονομική και κοινωνική, ε, και στην Επιτροπή Περιφερειών να μην κάνουν παράλληλους μονολόγους. Δηλαδή, θα πρέπει να συνεννοούνται πολύ περισσότερο και τα όργανα αυτά όταν γνωμοδοτούν για κάποια νομοθεσία. Να υπάρχει καλύτερο συντονισμός και για τον Λόρδο Μπόσουελ, Πρόεδρε, θα πρέπει να απαντηθεί η ερώτηση αυτή, το μεσημέρι κατά τη διάρκεια του γεύματος. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σάρλ Κέραντς έχει το λόγο. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ να σεβαστείτε το όριο των τριών λεπτών. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε διαφορετικά. Μην ξεπερνάτε τα τρία λεπτά. Ο Σάρλ σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προσυπογράφω και με τα δύο χέρια αυτά που είπαν οι δύο συνεισηγητές, η κυρία Μπρέσο και ο, ο κύριος Μπρόκ για τις ευκαιρίες που θα πρέπει να δράξει τόσο το Ευρωπαϊκό όσο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Εγώ θέλω να είμαι εξαιρετικά συγκεκριμένο στη δική μου πρόταση. Εδώ και χρόνια, είτε ως βουλευτής του Εθνικού Κοινοβουλίου, είτε ως ευρωβουλευτής, συμμετέχω σε τέτοιου είδους διαδικασίες και συνεδριάσεις και πάντα κάνουμε τις ίδιες διαπιστώσεις. Πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα που γνωρίζει πάρα πολύ καλά και ο εκπρόσωπος τη Βουλής του Λουξεμβούργου, μια χώρα που γνωρίζω πολύ καλά κι εγώ. Αυτό είναι ο δημοκρατικός κοινοβουλευτικό έλεγχος και ε, ο ρόλος της πολιτικής όθηση που μπορούμε να διαδραματίσουμε όταν έχουμε συντρέχουσες αρμοδιότητες. Ένα παράδειγμα. Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Ανάπτυξης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει καθόλου λόγο για τον προπολογισμό του. Τα εθνικά κοινοβούλια που ελέγχουν τι κυβερνήσει του ελέγχουν ένα μικρό κλάσμα των επενδύσεων που κάνει το μικρό Ευρωπαϊκό Ταμείο επενδύσεις ε, Ανάπτυξης και ο έλεγχος είναι στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι εκτελεστικό όργανο. Και τελικά κανείς δεν ελέγχει. Υπάρχει κανένα εθνικό κοινοβούλιο που να ελέγχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, ετησίως. Αυτό δεν θα ήταν στοιχειώδες. Επίσης, η συνθήκη της Λισαβόνας ορίζει ότι οι πολιτικές, εθνικές και ευρωπαϊκές στην αναπτυξιακή συνεργασία θα πρέπει να συντονίζονται καλύτερα και να είναι πιο συνεκτικές. Αυτό είναι υποχρεωτικό. Ποιο ασχολείται με αυτά τα θέματα σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Εγώ θα πρότεινα να επιφορτήσουμε δύο τρία πρόσωπα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δύο-τρεις από τα Εθνικά Κοινοβούλια για να συνεννοηθούν και να καταλήξουν σε μία μέθοδο έτσι ώστε να ε, ελέγχουμε αλλά και να προτείνουμε ε, από πλευρά των 29 ε, κοινοβουλίων όπου 29 ίσον 28 εθνικά συνένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να έχουν λόγο και τα κοινοβούλια, τα οποία κάνουν κοινοβουλευτικό έλεγχο, ε, κάνουν νομοθετική ε, δουλειά και νομοθετικές προτάσεις και πολιτικές. Θα παρακαλούσα λοιπόν την κυρία Πρέσο και τον Έλμαρ Μπρόκ να μας απαντήσουν. Πώς τη βλέπετε αυτή την πρόταση, να αναλάβει την πρωτοβουλία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να έχουμε κάθε χρόνο κοινέ συνεδριάσεις τέτοιου τύπου για θέματα που εκφεύγουν του γνήσιου κοινοβουλευτικού ελέγχου. Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα και Είναι πραγματικά μπαρόκ καμιά φορά οι μηχανισμοί λήψης αποφάσεων. Στην αναπτυξιακή συνεργασία με τρίτες χώρες. Και δεν απαγορεύεται πουθενά από τις σημερινές συνθήκες κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ. Σάγλα. Η Αρ... Αρμίνα Σπλιντέκ από τη Λιθουανία. Ε, yeah. Merci, Madame Présidente, chers collègues, chers amis. Pour moi, très difficile parler français, je préfère lituanien. Α, τελικά αποφάσισα να μιλήσω τη Λιθουανική. τα κοινοβούλια των κρατών μελών επιθυμούν η φωνή τους να ακουστεί. Ο πολιτικός διάλογος τον οποίο είχαμε μέχρι σήμερα με τα ευρωπαϊκά όργανα δεν είναι επαρκής. Ο διάλογος θα πρέπει να διευρυνθεί, θα πρέπει να βρούμε νέα μέσα τα οποία θα ενθαρρύνουν την πιο ενεργή συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Όλα αυτά μπορεί να γίνουν επί τη βάση των ισχυουσών συνθήκων. Πρέπει να αναπτύξουμε λοιπόν τον πολιτικό διάλογο προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, θα πρέπει εμείς να διευρύνουμε τον πολυμερή διάλογο ανάμεσα στα Κοινοβούλια και την Επιτροπή. Δεύτερον, θα πρέπει να αναπτύξουμε τον πολιτικό διάλογο ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι εννοώ όταν αναφέρομαι σε πολυμερή διάλογο. Μιλάω για μια συλλογική προσπάθεια διαλόγου των κοινοβουλίων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια από τις νέες ιδέες τις οποίες έχουμε προτείνει και μία από τις ιδέες τις οποίες θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε κατά τη διάρκεια της ε, Λιθουανικής Προεδρίας στο Συμβούλιο, το είχαμε θέσει τότε, ήταν τα συμπεράσματα τα οποία είχαν γίνει δεκτά στα πλαίσια της συνάντησης των Προέδρων των Κοινοβουλίων. Και νομίζω ότι τα συμπεράσματα αυτά είχαν αποσταλεί τότε στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο. Τα συμπεράσματα λοιπόν στα οποία είχαμε καταλήξει κατά τη διάρκεια της Λιθουανής Προεδρίας στην ουσία εκφράζουν τις απόψεις συλλογικά των κοινοβουλίων των κρατών μελών. Οι απόψεις τους είναι καθοριστικός νομίζω παράγοντας έτσι ώστε να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις γύρω από τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις πρωτοβουλίες φυσικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει σημασία να τα συζητήσουμε όλα αυτά από κοινού σε συνεργασία με τους εκπροσώπους λοιπόν της Επιτροπής και τους εκπροσώπους των κοινοβουλίων των κρατών μελών. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων και σε γραπτό επίπεδο και φοβάμαι ότι ο συντονισμός βέβαια που θα οδηγήσει σε μια τέτοια μορφή συνεργασίας δεν είναι εύκολος, αλλά είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη κοινοβουλευτική εμπλοκή. θα πρέπει να υπάρξει μια ξεκάθαρη ευρωπαϊκή πολιτική σε κοινοβουλευτικό επίπεδο η πολιτική αυτή που θα εμπλέκει τα κοινοβούλια των κρατών μελών μπορεί να ωφεληθεί και από τον μηχανισμό της πράσινης κάρτας. Και νομίζω επίσης ότι και η Κοζάκ είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία ε, χρήσης ε, ε, αυτής της μορφής συνεργασίας. Νομίζω ότι τα κοινοβούλια των κρατών μελών δεν θέλουν να ανταγωνιστούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά οι προτάσεις οι οποίες προέρχονται από τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι να καταστεί εφικτό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κατανοήσει πλήρως τις προσδοκίες των κρατών μελών. Ο κύριος Κουτσουπτσάν από τη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τα μέλη σας για την πρόσκληση σε αυτή την πραγματικά επίκαιρη συνάντηση. Πιστεύουμε πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεργάζεται όχι μόνο με τα εθνικά κοινοβούλια των ε, κρατών μελών αλλά και των υποψήφιων προς ένταξη χωρών. Γι' αυτό λοιπόν ε, μας ευχαριστεί πάρα πολύ η πρόσκλησή σας και με χαρά μέσα αναμένουμε και μελλοντικέ προσκλήσεις ε, σε παρόμοιες συναντήσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις και για να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια και τις προκλήσεις η Τουρκία πιστεύουμε πως ε, μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν ε, ασφάλεια, καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την διαχείριση της ε, προσφυγικής κρίσης. Φαίνεται πως το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα στηριχτεί στα εξή δύο θέματα. Καταρχάς σε εσωτερικά ζητήματα, με τα 500 ε, εκατομμύρια πολιτών που ζουν στα μέχρι τώρα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ανησυχίες, οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των πολιτών. Είναι ζωτική σημασία σε αυτό και ο, δεύτερο τα εξωτερικά ζητήματα, τα οποία είναι πιο επίκαιρα και πιο σημαντικά από ποτέ. Και θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω τα, ότι εμείς καταδικάζουμε φυσικά τα τραγικά γεγονότα στο Παρίσι. Και ας μην ξεχνάτε ότι τον Οκτώβριο είχαμε πολλά θύματα σε παρόμοια τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα και επίσης είχαμε και τις επιθέσεις στη Βηρητό. Θέλουμε λοιπόν να εκφράσουμε την ε, στήριξή μας και ε, σε αυτούς ε, τους λαούς. Πιστεύουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με την Τουρκία διότι αυτό είναι προς όφελος ε, όλων δεδομένων των καιρών ε, που ζούμε. Πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταφέρει να ξεπεράσει αρκετά προβλήματα εμβαθύνοντας την ε, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά και μέσω της διεύρυνσης. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι η στήριξη όχι μόνο των Εθνικών Κοινοβουλίων αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην Τουρκία είναι ε, πάρα πολύ ε, καλή. Την 1η Νοεμβρίου είχαμε εκλογές, έχουμε μια νέα κυβέρνηση και πιστεύω πως η νέα κυβέρνηση αυτή θα καταβάλει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες για να επιταχύνει την ε, ενταξιακή διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω λοιπόν πως πρέπει να δούμε αυτά τα πράγματα με πιο επικοδομητική και θετική ματιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργο Λάινεν τώρα έχει το, έχει το λόγο από τους Σοσιαλδημοκράτες. Ευρωβουλευτή. Σα ευχαριστώ πολύ, αγαπητή κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι έχουμε ευθύνη για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Κάθε ένα από εμά με το δικό του τρόπο και με τι ειδικέ του δυνατότητε είναι εκπρόσωπος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς ως εκπρόσωποι των πολιτών έχουμε ιδιαίτερη ευθύνη. Έχουμε ευθύνη για 550 εκατομμύρια πολίτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο-τρία σημεία και να πω καταρχάς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ε, επιτρεπεί να κατακαιρματιστεί. Στην Επιτροπή ΑΦΚΟ πήγαμε στο Λονδίνο και αυτά που ακούσαμε μας δημιούργησαν πάρα πολλές ε, σκέψεις ε, διότι δεν είδαμε ότι πρόκειται για μια Ευρώπη ενωμένη. Υπάρχει μια Ευρώπη, ούτε καν πολλών ταχυτήτων. Υπάρχει μια Ευρώπη αλακάρτο. Ο καθένα κάνει ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να επιλέξει ε, τι θα ακολουθήσει και τι όχι. Αυτό έχει αλλοιώσει τον χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κινδυνεύει να τον καταστρέψει. Και πρέπει λοιπόν να αναδώσουμε μεγάλη προσοχή στο να μην γίνει αυτό. Αυτό φαίνεται τώρα με την προσφυγική κρίση και με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Φαίνεται ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη το κάθε κράτος μέλο μόνος του δεν είναι αρκετά δυνατό για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε αυτόν τον συλλογικό χαρακτήρα και να μην ε, είμαστε απομονωμένοι στις ενέργειές μας. Γι' αυτό χρειάζεται όμως και περισσότερη διαφάνεια και περισσότερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, όσον αφορά το πόσο μπορεί να συμπεριληφθεί περισσότερο το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, ε, να σας πω πως αυτό είναι ένα πρόβλημα που μας απασχολεί πάρα πολύ καιρό. Υπάρχει ένα πρόβλημα καταρχάς ε, ταχύτητα στην επεξεργασία των θεμάτων και χρειάζεται καλύτερος συντονισμός. Ορισμένοι μάλιστα έχουν προτείνει και μία κοινή συνεδρίαση Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων έτσι ώστε να συντονιστούμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή. Χρειάζεται λοιπόν πολύ καλή συνεργασία και καλή πληροφόρηση. Τώρα, το ζήτημα της κίτρινης κάρτας είναι ένα μέσο το οποίο έχω την εντύπωση ότι είναι κάπως αμυντικό. Η κίτρινη κάρτα είναι τρόπον την ένα μέσο άμυνας το οποίο δεν μπορεί να είναι φυσικά ως τέτοιο αρκετά αποτελεσματικό. Πολύ... Για πολύ καιρό προσπαθήσαμε στα πλαίσια της ΕΚΟΣΑΚ να δώσουμε μια λύση και βλέπουμε ότι και άλλα κοινοβούλια έχουν ζητήσει στήριξη για κάτι που εγώ βρίσκω αρκετά αμυντικό όπως σας είπα. Ε, φυσικά υπάρχει και μια θετική εξέλιξη και αυτή είναι η πράσινη κάρτα που μας δείχνει τη θετική ε, πλευρά της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και σωστά αναφέρθηκε και ο Λόρδος Μπόσουελ σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μονοπόλιο στο δικαίωμα πρωτοβουλίας. Ούτε εμείς ούτε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμμετέχουμε σε αυτό και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να επανεξετάσουμε το θέμα και να συζητήσουμε διοργανικά για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τροποποιήσουμε το θεσμικό πλαίσιο. Διότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, επικρατεί μια δυσπιστία προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο καθένας ε, δεν εμπιστεύεται τον εταίρο του, γι' αυτό λοιπόν πρέπει, πιστεύω, να το εξετάσουμε. Σας ευχαριστώ. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Η Άννα Πίρτσα από το Κοινοβούλιο της Ρουμανίας έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να σας συγχαρώ που οργανώσατε αυτή τη συνάντηση σε μια πάρα πολύ επίκαιρη στιγμή. Είναι προφανές ότι έχουμε μπροστά μας μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη διεθνή σκηνή. Μετά από τις τρομοκρατικές ενέργειες στο Παρίσι, βλέπουμε να προστίθενται περαιτέρω κρίσεις οι οποίες σωρεύονται τελικά τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση επίσης της αντιευρωπαϊκής ρητορικής, η ελληνική κρίση, το μεταναστευτικό, ο Συριακός εμφύλιος και οι τρομοκρατικές ενέργειες. Απαιτείται λοιπόν να στρέψουμε την προσοχή μας σε μια προσπάθεια κοινών απαντήσεων στις σημερινές προκλήσεις. Μετά από χρόνια συζήτησης και διαπραγματεύσεων βλέπουμε ότι τα αντιευρωπαϊκά ε, κινήματα έπεισαν ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η ίδια η Ένωση φταίει για πάρα πολλές από τις αποτυχίες και από τα προβλήματα. Η συνταγματική συνθήκη ε, δεν ήθελε να υποκαταστήσει τα συντάγματα των κρατών μελών, κάτι το οποίο έτσι και αλλιώ είναι πολύ μακριά από τη σημερινή πραγματικότητα γιατί τα διάφορα κράτη-μέλη δεν θέλουν να συζητήσουν καν τα πλεονεκτήματα μιας πολυνικής ένωσης. Αυτό δεν επιτρέπει την περαιτέρω εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό ακριβώς έχει χάσει την εμπιστοσύνη και την αυτοεκτίμησή της. Μερικές φορές υφίσταται και κρίσεις τις οποίες αντιμετωπίζει εκτός νομικού πλαισίου, θέτοντας όμως θέματα δημοκρατικής νομιμότητας. Για να υπάρξει μια ακόμα πιο στενή συνεργασία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να ληφθούν υπόψη οι προσδοκίες οι οποίες υπάρχουν και μόνο τότε θα αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές προκλήσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει ότι η αδίποτε περαιτέρω αλλαγή σε επίπεδο συνθήκης θα πρέπει να συνοδευτεί από αλλαγές σε επίπεδο συνταγματικό. Ελπίζω οι μελλοντικέ ενέργειες που θα αναλυφθούν λόγω ακριβώς της ύπαρξης της πολιτικής βούλησης θα είναι αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν με διαφρομένο τρόπο και όχι ε, με αυθαίρετες ερμηνείες. Λόγω των μεταναστευτικών προβλημάτων τώρα τίθεται το θέμα της διακοπής ισχύω της συνθήκης Σέγγεν. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες τώρα, γιατί γνωρίζετε πόσο άδικο είναι για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία να μην έχουν ενταχθεί στο Σέγγεν, ενώ η Ρουμανία λειτουργεί όπως είναι κανονικά τα de μέλη, υπερασπιζόμενη το δεύτερο μεγαλύτερο εξωτερικό σύνορο και από ό,τι φαίνεται το κάνουμε καλά σύμφωνα με την έκθεση της Frontex. Η Ρουμανία παρέχει σταθερότητα και ασφάλεια για μια ευαίσθητη περιοχή για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Να υπογραμμίσω όμως ότι το Σέγγεν είναι ένα από τα πιο επιτυχή παραδείγματα ενισχυμένης συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό <clears throat> η ε, Ρουμανία θεωρεί ότι θα πρέπει το κεκτημένο αυτό να γίνει αντικείμενο προστασίας και να μην περιοριστεί η ελευθερία διακίνησης. Απαιτούνται αλλαγές στο εσωτερικό της Ένωσης, αλλαγές όμως οι οποίες να είναι ασεμβατές με τις αρχές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και γι' αυτό η Επιτροπή μου θα συνεχίσει να στηρίζει τους στόχους της ενίσχυσης της πολιτικής συνεργασίας δίδοντας εγγυήσει ε, για μη διακριτική μεταχείριση, για σεβασμό των θεμελιωδών αξιών, στηρίζοντας επίσης ε, και το streamlining της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων. Ας ελπίσουμε ότι από την παρούσα κρίση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βγουν ισχυρότερες και όχι με περισσότερες από τις σήμερα διαιρέσεις. Συνεπώς λοιπόν ε, ζητάμε, απευθύνουμε έκκληση έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή με ενωτικό τρόπο. Από την κάμερα dei deputati. Ο Ανδρέα Ματιώτη. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσπάθεια. Νομίζω ότι τέτοιου είδους επαφές θα πρέπει να είναι πιο συχνές όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι, η εποχή είναι διαφορετική από τις προηγούμενες. Ακόμα και η οικονομική κρίση ήταν κάτι το διαφορετικό από την σημερινή. Η σημερινή κρίση έχει σχέση με τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές των κοινωνιών μας. Γι' αυτό λοιπόν στην παρούσα φάση η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να παίξει ένα σημαντικό ρόλο θα συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπε ο κύριο Σανζέλ, ότι δηλαδή το θέμα της δημοκρατίας ή της έλλειψης δημοκρατίας είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιούμε με υπερβολικό τρόπο. Το πρόβλημα είναι η απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στα θεσμικά όργανα με τους πολίτες και με τα κοινοβούλια τα εθνικά. Η δική μου εμπειρία λέγει ότι η προσοχή την οποία δίδουν τα τοπικά κοινοβούλια και οι πολίτες <clears throat> στην νομοθετική δραστηριότητα και στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιστοιχεί στην σημασία των τεκτενομένων. Πάρα πολύ συχνά η συζήτηση αυτή θεωρείται ε, σαν μια μορφή επικοινωνίας ανάμεσα στην Ευρώπη και μια συγκεκριμένη χώρα και όχι σαν ένα ευρύτερο πολιτικό θέμα και αυτό αλλοιώνει τη σχέση της συνεργασίας. Οι περισσότερες νομοθετικές ρυθμίσεις που κυβερνούν τις χώρες μας προέρχονται από την Ευρώπη. Κι όμως η αντίληψη αυτή, η λογική αυτή δεν θεωρείται μια κοινή διαδικασία ανάμεσα στα κοινοβούλια και τις ευρωπαϊκές αρχές, αλλά σαν μια αντιπαράθεση ανάμεσα στα κοινοβούλια και την Ευρώπη. Και αυτό επηρεάζει τη σχέση με τους μεμονωμένους πολίτες. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας. Έγιναν πολλά σχόλια σήμερα στις θεσμικές αλλαγές και στις αλλαγές ανάμεσα στις, για τις σχέσεις των ε, οργάνων. Και οι προτάσεις Μπρέσο και Μπρόκ είναι θετικές. Το μόνο που θα μπορούσα να προσθέσω και δεν χρειάζεται να επανέλθω γιατί τα θέματα αυτά τα παρουσίασαν πολύ σωστά είναι η φυσική παρουσία του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις σχέσεις τους με τα κοινοβούλια. Ξέρω ότι ο κύριος Τίμερμαντς είπε ότι θα υπάρξει μια ισχυρότερη παρουσία της Επιτροπής και του α, Κοινοβουλίου. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη όχι μόνο σε σχέση με τα πολιτικά κόμματα, αλλά γενικότερα να δούμε ποια είναι τα συγκεκριμένα θέματα τα οποία πρέπει να τεθούν αυτή τη στιγμή σε συζήτηση και τα οποία θα πρέπει να γνωστοποιηθούν προς το κοινό και όχι μόνο στα μέλη των κοινοβουλίων. Στο κοινό, στα μέσα ενημέρωσης έτσι ώστε να γνωρίζουν τι συζητάμε. Η γνώση αυτών των θεμάτων δεν είναι σαφή σήμερα. Η άποψη είναι ότι τα θέματα αυτά επιβάλλονται εκ των άνω ενώ πολλές φορές ε, οι κυβερνήσεις μας συμμετέχουν και οι αποφάσεις είναι καρπός της συγκεκριμένη συμμετοχής. Ευχαριστώ πολύ από την Ουγγαρία και την Εθνοσυνέλευση, ο κύριος Μάτιας Φίλς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, κύριε Υπουργέ. Συμφωνούμε όλοι στη διαπίστωση ότι από τη θέση ισχύ της ε, συνθήκης της Λισαβόνας δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που μας παρέχει η συνθήκη αυτή. Τα εθνικά κοινοβούλια έχουν αρχίσει κάπως να προβληματίζονται για να δουν πώς ε, ε, θα μπορέσουν να συνεργαστούν καλύτερα. Θα πρέπει να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις ε, έχει αρχίσει αυτή η συνεργασία και οπωσδήποτε ε, η συνεργασία αυτή θα πρέπει να γίνει εντός των συνθήκων. Το είπε και ο κύριος Μπρόκ, δεν χρειάζεται τροποποίηση της συνθήκης. Ενισχυμένος λοιπόν διάλογος, έχουμε τη διαδικασία της πράσινης κάρτας πλέον και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βελτιωθεί και ο μηχανισμός της κίτρινης κάρτας. Όλα αυτά έχουν συζητηθεί, έχουν γίνει προτάσεις, τα είπαν και οι προλαλήσαντες. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να εκμεταλλευτούμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Καλές είναι οι νέες προτάσεις και συζητήσεις που γίνονται, αλλά θα πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη τα υφιστάμενα μέσα. Διαθέτουν δυνατότητες τα Εθνικά Κοινοβούλια και πρέπει να βελτιωθούν οι διαδικασίες. Έχουμε δυνατότητες τις οποίες δεν αξιοποιούμε 100% εθνικά κοινοβούλια εκπροσωπούν τους Ευρωπαίους πολίτες και εξασφαλίζουν την ε, επικοινωνία με τους πολίτες και την επαφή τους με όλες αυτές τις ευρωπαϊκές διαδικασίες. Βουλευτές, γερουσιαστές των Εθνικών Κοινοβουλίων προφανώς βρίσκονται πιο κοντά στους πολίτες και είναι πιο εύκολο εμείς να ε, ε, τους μεταφέρουμε και να τους διαβιβάζουμε τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Το σημείο 9 του εγγράφου εργασίας έχει ένα ενδιαφέρον. Να συνεργάζονται λοιπόν καλύτερα οι ε, Ευρωπαϊκές Κοινοβουλευτικές Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις ε, εκάστοτε εθνικές. Θα πρέπει να υπάρχουν ε, ειδικέ προτάσεις ε, όμως ε, για να αντιμετωπίσουμε και τρέχοντα προβλήματα όπως είναι το προσφυγικό, το μεταναστευτικό, η συνεργασία στην άμυνα και η συνεργασία με το ΝΑΤΟ, που καλό θα ήταν να ενισχυθεί. Γίνεται λόγος για τρίτες χώρες ε, που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση που δεν είναι ασφαλής. Θα πρέπει να ληφθεί ε, μια απόφαση ε, σχετικά με το τι γίνεται με τη διαδικασία ασύλου. Τι λέει η Ουγγρική Βουλή. Είναι πολύ καλό αυτό το έγγραφο εργασία ως βάση όμως και αφετηρία για μια συζήτηση και αν ε, προχωρήσουμε στην κατεύθυνση αυτή χωρίς αναθεώρηση των συνθηκών μπορεί να βελτιωθεί η συμμετοχή των κοινοβουλίων προς όφελος όλων των κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ. Um, Αγαπητοί συνάδελφοι, εξαλείφθηκε εδώ ο κατάλογος των ομιλητών. Ε, οπότε θα δώσουμε ξανά το λόγο στην κυρία Μπρέσο ε, και μετά στον Υπουργό για να δευτερολογήσουν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν έχω το χρόνο για να μπω στην ουσία των πολλαπλών παρατηρήσεων οι οποίες προηγήθηκαν. Πάντως ε, τις λαμβάνουμε υπόψη και θα ήμουν ευγνώμων προς όλα τα κοινοβούλια των κρατών μελών να μας αποστείλουν αν είναι δυνατόν και τα γραπτά του κείμενα έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη ηρεμία. Λίγα πράγματα θα ήθελα να τονίσω. Πρώτον, στο βασικό θέμα την προσπάθεια δηλαδή α, ανείχνευσης των δυνατοτήτων της συνθήκης της Λισαβόνας υπάρχει μια σαφής συνένεση και αυτό το εκτιμώ δεόντως γιατί πάρα πολλές φορές έχουν υπάρξει αιτήματα εμβάθυνσης ορισμένων θεμάτων στα πλαίσια της συνθήκης. Αυτό θα το κάνουμε. Νομίζω ότι φάνηκε με ξεκάθαρο τρόπο ότι είναι σημαντικός ο ρόλος τον οποίο καλούνται να παίξουν τα εθνικά κοινοβούλια στην νομική και πολιτική διαδικασία στην Ευρώπη. Νομίζω ότι αν πράγματι θέλουμε εμείς να περάσουμε σε περαιτέρω πολιτική και οικονομική ολοκλήρωση, υπάρχουν θέματα τα οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Η καλύτερη σχέση ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα τα νομοθετικά θα μπορέσει να βοηθήσει την πολυεπίπεδη αν θέλετε διακυβέρνηση. Ξέρετε ότι και η Περιφερειακή Επιτροπή το επιθυμεί αυτό είναι τόσο περίπλοκη η Ήπειρος μας, είναι τόσο πολλαπλές οι αντιπροσωπευτικές οργανικές δομές, δημοκρατικές όλες, αλλά με διαφορετικά ιστορικά στοιχεία, με διαφορετικά πολιτιστικά στοιχεία. Και σχετικά τώρα με τις διάφορες πολύχρωμες κάρτες στις οποίες αναφερθήκατε. Νομίζω ότι θα πρέπει να μείνουμε ε, μέσα στη συνθήκη βασικά γιατί το τι μπορεί να συμβεί εκτός των συνθήκων, εκτός θα δούμε. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε στο εσωτερικό της συνθήκης της Λισαβόνας να ορίσουμε μία διαδικασία η οποία να είναι προϊόν συμφωνίας ανάμεσα στο Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως και τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων να προβλεφθεί μια διαδικασία λοιπόν η οποία θα μας επιτρέψει έστω και σε μια πρώτη φάση πειραματική να βρούμε την σωστή μέθοδο συνεργασίας. Η συνεργασία αυτή δεν θα έχει σαν στόχο μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Συμβούλιο. Και τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εκπρόσωπο του Τουρκικού Κοινοβουλίου Πρώτον για την παρουσία του είναι σημαντική. Οι χώρες οι οποίες έχουν εμπλακεί στη διαδικασία ένταξης να συμμετέχουν στις συζητήσεις μας. Και σε ό,τι με αφορά, ε, και νομίζω ότι αυτό ισχύει για όλους, ελπίζω να συνεχιστεί ο διάλογος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για να αντιμετωπίσουμε τις κοινέ απειλές η συνεισφορά και της δικής τους χώρας θα είναι κομβική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Ντανούτα που μου έδωσε ε, το λόγο. Να πω πολύ σύντομα ότι υπάρχει μεγάλη συνένεση ε, για το ότι δεν πρέπει να αγγίξουμε τις συνθήκες. Ε, για δύο λόγους, όχι μόνο επειδή θα ανοίξουμε το κούτι της Πανδώρας, αλλά και επειδή ακόμα μπορούμε εντό των συνθήκων να κάνουμε πάρα πολλά. Μας επιτρέπουν πολλά οι συνθήκες και η κυρία Μπρέσο και ο κυρίος Μπρόκ με τις παρεμβάσεις τους μας έδωσαν πολλά παραδείγματα, καθώς και άλλοι συνάδελφοι, για το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Να επανέλθω και να πω κάτι που δεν είπα πιο πριν. Υπάρχουν κάποιες εξειδικευμένες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες πιστεύω πως θα έπρεπε να έχουν καλύτερη συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια. Και να σας πω ότι στα εθνικά κοινοβούλια συνήθως δημιουργείται μια ευρωπαϊκή ελίτ. Γι' αυτό λοιπόν ε, πρέπει να προσπαθήσουμε ώστε κάθε μέλος ενός εθνικού κοινοβουλίου να ε, προσθέτει και την ευρωπαϊκή διάσταση πέρα από την ε, τοπική, την περιφερειακή και την εθνική. Χρειάζεται λοιπόν να σταματήσουμε να δημιουργούμε αυτές τις ευρωπαϊκές ελίτ, αλλά να φέρνουμε την ευρωπαϊκή διάσταση σε όλες τις επιτροπές. Γι' αυτό λοιπόν με χαροποίησε ιδιαίτερα η πρόταση του Σάρλ Γκέρενς για να υπάρχουν δηλαδή κοινέ αρμοδιότητες έτσι ώστε να μπορούμε να συντονιζόμαστε καλύτερα. Για παράδειγμα με το Ταμείο ε, ανάπτυξης, όπως και η πρόταση του κυρίου Λάινεν που μας είπε πως χρειάζεται καλύτερη ε, συνεργασία, καλύτερο συγχρονισμός και πως θα μπορούσε να υπάρχει επίσης ε, μία εβδομάδα κατά την οποία θα μπορούμε να συζητήσουμε το ετήσιο πρόγραμμα ε, του κάθε κοινοβουλίου. Πιστεύω πως αυτές είναι προτάσεις προς την σωστή κατεύθυνση. Τέλος, να πω ότι στην Κόσακ είχαμε μία μεγάλη συζήτηση για την πράσινη κάρτα που δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και Αναρωτιόμασταν μάλιστα στην αρχή αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον όρο πράσινη κάρτα ή τον ενισχυμένο πολιτικό διάλογο. Προτιμήσαμε το τελευταίο διότι θέλαμε να υπάρχει ένας ε, πραγματικό διάλογος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε καταρχάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά να καλέσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να καταρτήσει μία λευκή ή πράσινη βίβλο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ε, έτσι έχουν τα πράγματα στην ΚΟΣΑΚ. Του των λεξέντων ε, να σας πω ξανά ότι χάρηκα πάρα πολύ για τη διοργάνωση αυτής της συνάντησης και ε, ανυπομονώ να ακούσω το, τους συμμετέχοντες το απόγευμα. Να σας συγχαρώ λοιπόν ε, σας, την Επιτροπή σας, η συνεισφορά σας είναι πάρα πολύ σημαντική και στην Κόσακ να σας πω πως υπάρχει πάρα πολύ θετικό κλίμα και ανυπομονούμε όλοι να συνεργαστούμε μαζί σας τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Μάρκ. Θα ήθελα και εγώ πριν διακόψουμε να πω ότι καταρχάς είναι και για μας σημαντικό. Υπάρχουν πολλές πλατφόρμες συνεργασίας ε, ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά με αυτήν την ε, συνεδρίαση δημιουργούμε και ε, μια πλατφόρμα για άλλα θέματα τα οποία είναι πολύ προσφυλή σε εμά και μάλιστα εμπίπτουν και στις αρμοδιότητές μας. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν. Ήταν η αρχή, ήταν τα πρώτα βήματα για μια καλή συνέχεια. Και να σας πω, Λόρδε Μπόσουελ, ότι σίγουρα θα ε, δώσουμε μεγάλη προσοχή στην επιστολή σας και να είστε σίγουρος πως δεν πρόκειται να την αγνοήσουμε. Λοιπόν, ε, στην αίθουσα νούμερο 4, το σαλόν νούμερο 4 είναι στο ισόγειο δεξιά. Όπου βρίσκονται και τα άλλα εστιατόρια. Θα τα πούμε εκεί. Ευχαριστώ.